Good afternoon and welcome. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στην ε, απογευματινή συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ο πρόεδρος ο Ζων Χτουί θα έρθει από τις 4 και μου ζήτησε να προεδρεύσω στην πρώτη αυτή φάση της πρώτης ώρας όπου θα συζητήσουμε το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως ξέρετε, έχουμε υιοθετήσει σήμερα το πρωί σε επίπεδο Επιτροπής ε, το ψήφισμα για το έγγραφο προβληματισμού που εκδόθηκε από την Κομισιόν για το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κ. Γιάνν Όλμπριχτ και η κυρία Ιζαμπέλ Τομάη, δύο εισηγητές μας, θα ετοιμάσουν μια έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί και θα ψηφιστεί εδώ στις αρχές του 2018. Ούτως ή άλλως πριν προτείνει η Κομισιόν τη θέση της που θα το κάνει το Μάιο. Ο Γιάνν Λεβαντόσκι και ο Ζεάν Ντεπρέ, οι συγητές μας για τους ίδιους πόρους, ετοιμάζουν τη δική τους έκθεση, που θα παρουσιαστεί επίσης μέσα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ξεκινάμε τώρα ε, διάφορες συζητήσεις με εμπειρογνώμονες, όχι εντός του Κοινοβουλίου, εκτός του Κοινοβουλίου, και για τη σημερινή συνεδρίαση έχουμε την ε, συνάδελφο αυτή από το Αυτιακό Ινστιτούτο Ερευνών και τον κύριο Άρχοστ από το, Ιακωβίνου, από το Πανεπιστήμιο Ιακωβίνους της Βουδαπέστης. Αποφασίστηκε να οργανωθούμε ω εξή τι σημερινέ συζητήσει σε δύο τμήματα. Καταρχάς, για την δομή του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, όπου η κυρία Σράτσεν Στόλερ θα μιλήσει για αυτό το κομμάτι και ο άλλος συνάδελφος για το επόμενο θέμα που θα είναι η διάρκεια του πουδουπού. Πριν περάσουμε στα δύο αυτά σημεία, η δομή τη δομή δηλαδή και το, τη διάρκεια. Θα μας κάνουν κάποια εισαγωγικά σχόλια η κυρία Τομά και ο κύριος Όλμπριχτ. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. ορίζω τους εμπειρογνώμονες. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί τους την άποψή τους. Να υπενθυμίσω απλώς στους συναδέλφους ότι έχω μια συγκεκριμένη ατζέντα για τις εργασίες μας, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είμαστε στη φάση προετοιμασίας του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και έχουμε τη Γενική Πολιτική Συμφωνία. Θα, θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τα πάντα πριν ολοκληρωθεί αυτή η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, Κομισιόν. Δεν ξέρω αν θα γίνει δυνατόν, αλλά αυτό είναι το, ο στόχος μας. Έχουμε μια πρόταση καταρχάς από την Κομισιόν ε, στα πλαίσια ενός πακέτου και μιας ε, λευκής βίβλου για το, τη μελλοντική χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένες προτάσεις για τον προϋπολογισμό. Σήμερα το πρωί ψηφίσαμε ένα ψήφισμα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών που θα περάσει τώρα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο στην επόμενη δομέλεια δηλαδή, του Οκτωβρίου ε, που αντιδράμε στην πρόταση της Κομισιόν. Δηλαδή, αντιδρούμε για τη μέθοδο, για την προσέγγιση που προτείνει η Κομισιόν, για τις βασικές προκλήσεις ε, που θεωρούμε ότι υπάρχουν. Είναι το έγγραφο το οποίο ψηφίσαμε σήμερα το πρωί. Τώρα ξεκινάμε τις προετοιμασίες για την έκθεση δίας πρωτοβουλίας. Και σε αυτή την έκθεση θα θέλαμε να είστε πιο συγκεκριμένοι και θα θέλαμε να ακούσουμε απόψεις από διάφορες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις τομεακές πολιτικές, όπως το χάρη την πολιτική συνοχή, ε, την γεωργική πολιτική, την ε, έρευνα και καινοτομία κτλ. Θα ετοιμάσουμε αυτή την έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας μέχρι το Μάρτιο, γιατί η Κομισιόν υποσχέθηκε να παρουσιάσει το προσχέδιο του επόμενου Πουδουπού το Μάιο. Σε αυτό το έγγραφο της, έκθεσης, της γνωμοδότησης Ιδία Πρωτοβουλία, και γι' αυτό η σημερινή συνεδρία είναι σημαντική, θα θέλαμε να συλλέξουμε τα βασικά στοιχεία τη συζήτηση που θα λάβουν χώρα, των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες. Και στην έκθεσή μα θα έχουμε την γενική προσέγγιση για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και το Πουδουπού. Στο πρώτο τμήμα θα θέλαμε ως Κοινοβούλιο να προτείνουμε κάποια πράγματα για τη δομή του προπολογισμού. Τον τρόπο δηλαδή που κατασκευάζουμε, που φτιάχνουμε τον προπολογισμό. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί σε επόμενου μήνες θα είναι αν θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι στον προπολογισμό. Χρειαζόμαστε να αλλάξουμε τη δομή του προπολογισμού. Είναι απαραίτητο να προσθέσουμε κάτι, είναι, κάτι να αλλάξουμε, είναι απαραίτητο να αλλάξουμε κάτι στη φιλοσοφία του προπολογισμού θα έχουμε νέες προκλήσεις. Και το θέμα είναι πώς θα τις εντάξουμε αυτές τις προκλήσεις μέσα στο σημερινό πλαίσιο του προπολογισμού. Μήπως χρειαζόμαστε αλλαγέ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και τις απόψεις των ειδικών. Είμαστε ευγνώμονε που θα ακούσουμε το, τα όσα μας πει ο πρώτος για την δομή του επόμενου πουδουπού και, του, και των ιδίων πόρων. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Κάτι που θα υπάρχει στην έκθεση Λεβαντόσκη και Ντεπρέ ε, και θα αφορά τους ίδιους πόρους. Είναι τμήμα του πακέτου. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, δεν έχουμε πάρει απόφαση και για τους ίδιους πόρους. Επομένως, η πρώτη ερώτηση είναι τι γίνεται με τη φιλοσοφία του Πουδουπού, τη δομή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να τη διορθώσουμε, την αλλάξουμε ή να αλλάξουμε απλώς α, τις ανθιπολεπτομέρειες. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Η διάρκεια. Δεν είναι μόνο τεχνικό ερώτημα αυτό, δεν είναι θέμα χρόνου μόνο. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας των πολιτικών. Η δημοσιονομική δομή μπορεί να είναι χρήσιμη προωθώντας διάφορες πολιτικές. Θα ακούσουμε για αυτό το θέμα ε, να μας το παρουσιάζει ο δεύτερος ε, εμπειρογνώμονας. Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο. Πέντε χρόνια, εφτά χρόνια, πέντε συν κάτι. Θα ήθελα να ακούσω τους εμπειρογνώμονες. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, ας πούμε, κάθε μιας από τις προτάσεις που έχουμε επιτάπητος. Συνοψίζω, λοιπόν. Θέλουμε να παρουσιάσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου το Μάρτιο και για να την έχουμε Πρέπει να έχουμε μια ε, πραγματογνωμοσύνη και κάποια στοιχεία εμπειρογνωμόνων για να φτιάξουμε, για να πάρουμε θέση. Αυτά εν ώψη της διαπραγμάτευσης που θα γίνει. Αυτά σας υπενθυμίζω την, το χρονοδιάγραμμα. Και αυτά που θα μας πούνε οι εμπειρογνώμονες, τι θέση έχουν στη δουλειά μας. Θα τα λάβουμε υπόψη μας και κάποια θα απεικονιστούν και στη θέση που θα παρουσιάσουμε το Μάρτιο. Η Ιζαμπέλ Τομά. Πολύ σύντομα. Γιατί ο Ιαν τα είπε σχεδόν όλα και με κάλυψε σχεδόν 100%. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή μου και τους συναδέλφους που μας επέτρεπαν σήμερα το πρωί να εξασφαλίσουμε πλατιά πλειοψηφία στο ψήφισμα αυτό. Είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά προαναγγέλει μία, αν όχι συνένεση, τουλάχιστον μία πλειοψηφία, του ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και είναι καλό σημείο αφετηρίας. Επίσης, όπως είπε και ο Ιαν, μιλάμε για μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας. την οποία επεξεργαζόμαστε, γιατί οι διάφορες επιτροπές ε, ετοίμασαν τη δική τους νομοδότηση. Ε, θα έχει δύο τμήματα αυτή η έκθεση η πρωτοβουλία. Ε, μία για τον προπολογισμό, δηλαδή με όλα αυτά τα θέματα τα οποία σας είπε ο Γιάνν και τα οποία συζητήσαμε σήμερα, δηλαδή τις δομή του προπολογισμού, του δημοσιονομικού πλαισίου. Το θέμα της δομής συνδέεται και με το πώς θα επιλύσουμε το πρόβλημα της διαφάνειας για τον προπολογισμό. Δηλαδή να τον διαβάζει κανείς και να καταλαβαίνει τι λέει και τι σχέση έχει ο προϋπολογισμός με τις πολιτικές. Και παράλληλα να έχει και την απαραίτητη ε, ευελιξία που δεν είχε που δεν την είχε παρκώ αυτό το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Επίση το θέμα τη διάρκεια, όπω υπόθηκε επίση. Και εκεί υπάρχουν ε, δύο στοιχεία που πρέπει να παντρέψουμε από τη μία τη δημοκρατική διάσταση, ότι δηλαδή αυτή η διάρκεια θα πρέπει να συνδέεται με την εντολή που παίρνει από τους εκλογείς στο Κοινοβούλιο, αλλά και η Κομισιόν, και από την άλλη να συνδυαστεί με τα διαφορετικά ταμεία, έτσι, η διάρκεια αυτή. Και να υπάρχει μία συνάφεια. Όλα αυτά είναι πράγματα που εκ πρώτη όψεως μπορούν να φαίνονται αντιφατικά. Όμως, εμείς θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και ξέχασα να, ξε... να ευχαριστώ και κάποιον άλλο για το σημερινό ψήφισμα. Και την γραμματεία της Επιτροπής Προπολογισμών και τους πολιτικούς συμβούλους που έκαναν θαυμάσια δουλειά. Θα τους χρειαστούμε όλο αυτό το καιρό, όλα αυτά τα, όλους αυτούς τους μήνες μπροστά, που είναι μπροστά μας, γιατί τώρα αρχίζει η πραγματική δουλειά με την έκθεση πρωτοβουλία όταν την ετοιμάσουμε και μετά με τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ Ιζαμπέλ και Ιαν που θέσατε το πλαίσιο για τις συζητήσεις μας και τώρα θα περάσουμε στους δύο μιλητές. Πριν του δώσω το λόγο, να τους πω τα εξή. Πρώτον, οτιδήποτε και αν πούν, δεν δεσμεύει την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεν είναι η άποψή της. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Εν συνεχεία θα δώσουμε το λόγο ξανά στους εισηγητές, στους κοιόδους εισηγητές, τους ε, συντάκτες νομοδοτήσεων των άλλων επιτροπών να είναι παρόντες και τέλος στους βουλευτές της Επιτροπής Προπολογισμών. Για την πρώτη συζήτηση για τη δομή, η κυρία Σράτσεν Στόλερ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή την ε, συνεδρίαση, σε αυτή την ενδιαφέρουσα χρονική συγκυρία. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να σας παρουσιάζω το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι η γενικότερη προσέγγιση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διαμορφωθεί αναλογώς με τις προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε πέρα του Brexit και των επιπτώσεων που θα έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις εκτός από αυτός, όπως είναι η γύρη για τη διεύρυνση, οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Αυτά φαίνονται και στην έκθεση συνοχής, υπάρχουν τα διαρθρωτικά και δομικά προβλήματα των χωρών του Νότου, η κλιματική αλλαγή, οι δημογραφικές αλλαγές, η ενεργειακή μετάβαση, μειωμένη, μειούμενη αλλά παρά όλα αυτά υψηλή ανεργία και κυρίως ανεργία των νέων, των νέων αυξημένη ανισότητα ως προς το εισόδημα και το πλούτο, εμένων κίνδυνος φτώχειας, και κρίση προσφυγική και μεταναστευτική. Ένα βασικό δίδαγμα λοιπόν που μπορούμε να αντλήσουμε από το υφιστάμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ότι η δομή του έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή δεν φτάνει για να ε, αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις ούτε από πλευράς εσόδων ούτε από πλευράς δαπανών. Πολύ λίγο συμβάλλει π.χ. στο στόχο αηφόρου ανάπτυξης και βιώσιμης ανάπτυξης στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έτσι, έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε τη στρατηγική για το 2020, την ατζέντα για το 2030 για την αηφόρο ανάπτυξη, αλλά και τη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή των παρουσίων, Παρισίων του 2015. Όλα αυτά χαρακτηρίζονται από μεγάλα κενά ως προς την αηφορία και στα, στις δαπάνες και στα έσοδα. Σήμερα θα μιλήσω κυρίως για τις δαπάνες. Θέλω όμως να τονίσω ότι και το σύστημα των ίδιων πόρων πρέπει να μεταρρυθμιστεί και αυτό είναι επίγον για να μπορέσει να γίνει βιώσιμο. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυσμείο να σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση των υφιστάμενων έλλειμματων στη δομή των δαπανών σε επίπεδο ένωσης. Υπάρχει μια κάποια αλλαγή δαπάνες προς τομεί που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μακροπρόθεσμη μείωση του μεριδίου της γεωργικής πολιτικής στις γενικότερε δαπάνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα πρασίνισμα εντό εισαγωγικών των γεωργικών δαπανών. Έχουμε μια κάποια αύξηση των δαπανών για έρευνα, τεχνολογία και νοτομία, ωστόσο πολύ λίγα δίδονται για τα δημόσια αγαθά και πολύ λίγη είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ως προς αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί project που δημιουργούν μόνο τοπική προστιθέμενη αξία. Και αυτό στηρίζεται στην προοπτική των κρατών μελών που προσπαθούν να αξιοποιήσουν στο ε, μέγιστο ε, σε τοπικό επίπεδο τις εισφορές που κάνουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παρά τις προκλήσεις, οι καθαρές χώρες που συνεισφέρουν καθαρά είναι όλο και πιο επιφυλακτικές πολιτικές θέλουν όλο και λιγότερο να συνεισφέρουν και οι πολίτες φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται πόσο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός επηρεάζει θετικά τη ζωή τους. Παρά λοιπόν αυτές τις αλλαγές και τις μεταστροφές της προτεραιότητες, το υφιστάμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο συνεχίζει να κυριαρχείται από την κοινή γεωργική πολιτική, σχεδόν 40% παρόλο που το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί και βαίνει μειούμενο. Δεύτερο μεγάλο, δεύτερος μεγάλος τομέας δαπανών είναι η πολιτική συνοχής. Περίπου το 1 τρίτο του συνόλου των δαπανών μας στοχεύει στη συνοχή και 13% αύξηση βέβαια, αλλά συνεχίζει να είναι λίγη η δαπάνη για την ανταγωνιστικότητα, για τις υποδομές. 2% ε, του προϋπολογισμού αφιερώνονται στην αναπτυξιακή βοήθεια, στο τακτικό προϋπολογισμό και έχουμε και 30 δις ευρώ που δίδονται στο Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο εκτός Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και 1% του προϋπολογισμού για δαπάνες που έχουν σχέση με το Σέγγεν, διαδικασίες ασύλου, μετανάστευσης, συνόρων και εσωτερικής ασφάλειας. Αυτά λοιπόν για το υφιστάμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ως προς τους στρατηγικούς προσανατολισμούς. Έτσι όπως έχει η δομή αυτή τη στιγμή μας δείχνει ότι υπάρχουν κενά στην βιωσιμότητά του. Οι δαπάνες για τη γεωργική πολιτική σήμερα διατηρούν την, τις υφιστάμενες δομές παραγωγής εντός πρώτου πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Μεγάλο μερίδιο των ενισχύσεων στη γεωργία δίδεται σε μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δίνει προτεραιότητα επομένως στη συμβατική γεωργία. Και ο δεύτερος πυλώνας της κοινή γεωργικής πολιτικής που έχει περισσότερο να κάνει με την αηφορία και που θα μπορούσε να στηρίξει ενεργά την βιολογική γεωργία ανέρχεται περίπου στο 1 τέταρτο των συνολικών γεωργικών δαπανών. Και αυτή είναι μια πρώτη παρατήρηση. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι παρά τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην κοινή γεωργική πολιτική τις τελευταίες δεκαετίες, η γεωργική πολιτική και οι δαπάνες οι γεωργικές συνεχίζουν να τείνουν να έχουν σε ε, προσωπικό και περιφερειακό αποτέλεσμα ε, αντίστροφο, πιστοδρομικό, regressive effect. Από εκεί και πέρα το Ταμείο Συνοχή και τα κονδύλια Συνοχή στοχεύουν ιδιαίτερα στα παραδοσιακά project υποδομών και πολύ συχνά απουσιάζει η προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρκετά πλούσιε, χώρε ε, μέλη ωφελούνται από τι γεωργικές ενισχύσεις και τις ενισχύσει για τι υποδομές για τη συνοχή. Τα κονδύλια δεν αφιερώνονται στου πιο φτωχού με απολύτως στόχο τρόπο και όλα αυτά υπάρχουν στην έκθεση για τη συνοχή που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτον, οι δαπάνες για την έρευνα που έχουν πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και στην ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα. Είναι πολύ χαμηλές. Και συγκριτικά έχουμε λίγες δαπάνες εάν ερμηνεύσουμε σωστά τους αριθμούς που υπάρχουν στην ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 20% των δαπανών του ορίζοντα 2020 σχετίζεται με έρευνα που έχει να κάνει με το κλίμα. Και όλα αυτά συγκριτικά με το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι καλύτερα. Τότε ήταν 10% αν δεν απατώμε. όλα αυτά υπολείπεται του στόχου που έχει συμφωνηθεί. Τέταρτη παρατήρηση. Πολύ λίγη και μικρή χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει αποφασιστικά στην αναπτυξιακή βοήθεια και στη συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια για το μετριασμό των συνεπειών της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Το 2016 το 2,51% του GNI, των ε, καθάριστου εθνικού εισοδήματο, αφιερώθηκε σε αυτό και αυτό υπολείπεται από το στόχο που είναι 7% του GNI. Μετά από αυτή τη σύντομη επισκόπηση της υφιστάμενης δομής των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς για τη φύση του επόμενου πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου Προφανώς η προσέγγιση μας και για το επόμενο ΠΔΠ θα εξαρτηθεί από το ποιο από τα πέντε σενάρια θα ακολουθηθεί έτσι όπως βρίσκονται στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στα μέση του 2017 η Επιτροπή διαγράφει τις επιπτώσεις κάθε ενός από τα πέντε αυτά σενάρια σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της πολιτικές για ε, τις δαπάνες στους διάφορους τίτλους, στους διάφορους τομείς. Αν ακολουθηθεί το σενάριο που ότι θα κάνουμε όλοι μαζί λιγότερα, τότε ε, μόνο δεν θα αλλάξει η δομή μεταξύ δαπανών και εσόδων. Για τα άλλα τέσσερα σενάρια πρέπει να αλλάξει η δομή μεταξύ δαπανών και εσόδων, πρέπει να κινηθούμε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και πρέπει να έχουμε νέες συμφωνίες για τους ίδιους πόρους, να έχουμε νέους ίδιους πόρους ή άλλους πόρους εισοδήματος εξετάζοντας τις ανεπάρκειες και τα ελλείμματα του υφιστάμενου προϋπολογισμού με το υφιστάμενο πολιτικό, θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα λοιπόν υπέρ των θεμελιωδών αλλαγών στον προϋπολογισμό με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανεξαρτήτως ε, του ποιο από τα σενάρια για τη μελλοντική ευρωπαϊκή ενοποίηση ολοκλήρωση θα ακολουθηθεί τελικά. Είτε μιλούμε για ταχύτητα, για βάθος, για κατεύθυνση, για συγκεκριμένη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είτε μιλούμε για το ύψος, τον όγκο, το μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, Ε, και ακόμα και αν διατηρηθεί ο προπολογισμό και θα πρέπει να διατηρηθεί για όλη τη διάρκεια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου του επόμενου, σε κάθε περίπτωση η δομή μεταξύ δαπανών και εσόδων, η διάρθρωση πρέπει να αλλάξει, να μεταστραφεί, να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στη δυναμική της οικονομίας ε, στην κοινωνική συμπερίληψη και στην αηφορία, στη βιωσιμότητα, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, με βάση ε, τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για το Brexit, με βάση το ότι οι συζητήσεις για τη μελλοντική ολοκλήρωση και ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε εμβρυϊκό στάδιο. Θα πρέπει και δεν θέλω πολύ να το αναφέρω αυτό το ζήτημα, γιατί ο συνάδελφος θα πάρει το λόγο αργότερα και να το παρουσιάσει για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, με αυτά τα δεδομένα που μόλις τώρα ανέφερα, από τη μία έχουμε μία περίοδο 5 συν 5, άρα μία δεκαετή περίοδο με ενδιάμεση αξιολόγηση και αναθεώρηση. Εκεί θα έχουμε μακροπρόθεσμη σταθερότητα των δαπανών, αλλά πρέπει να έχουμε και ισχυρές ρήτρες αναθεώρησης με σημαντικό βαθμό ευελιξία μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών δαπανών. Να μπορούμε εύκολα δηλαδή να μεταφέρουμε χρήματα από τον ένα τομέα στον άλλο, ειδικά εάν τα κράτη-μέλη δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν για τα θεμελιώδη του προϋπολογισμού μετά το 2020. Είδα αλλιώς, η συζήτηση θα ξαναξεκινήσει από το 2020 και μετά, αν δεν προεπιλευθεί κάτι τέτοιο. Έρχομαι τώρα στην δομή, στη διάρθρωση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θέλω να πω κάποια βασικά που πρέπει όλοι να τα ξέρουμε για να έχουμε δαπάνες που θα είναι στραμμένες προς την αηφορία, προς τη βιωσιμότητα. Σε γενικές γραμμές, οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνονται σε τοπής πολιτικής, όπου οι συντονισμένες δράσεις των κρατών μελών δεν είναι αρκετές. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν περισσότερες από μία χώρες, υπάρχουν κάποια ζητήματα όπου διακυβεύονται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και βεβαίως πρέπει να τηρούμε πάντοτε την αρχή της επικουρικότητας. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα να αξιολογήσει τα μέτρα και να ποσοτικοποιήσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Να ένα ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένα άλλο κριτήριο είναι κατά πόσο η δαπάνη έχει διασυνοριακό στοιχείο. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδου κριτήρια που μπορούν να αποφασιστούν. Και αν δεν μπορεί να τηρηθούν αυτά τα κριτήρια, τότε είναι καλύτερο το κάθε θέμα να εξεταστεί από το κράτος μέλος μόνο. Διότι δεν δημιουργείται ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Ευρωπαϊκή προσταθεμένη αξία θα υπάρξει αν εστιαστεί στην αηφορία, στη βιωσιμότητα σε πολλούς τομείς πολιτικής μπορεί να έχουμε προστιθέμενη αξία. Καταρχάς μειώνοντας τις γενικότερες δαπάνες για τη γεωργική πολιτική, πρασινίζοντας τις άμεσες πληρωμές τους ε, γεωργούς, τους αγρότες, το πρώτο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής και οι γεωργικές δαπάνες να μεταστραφούν, να αλλάξουν, να πάνε στο δεύτερο πυλώνα, προκειμένου να σέβονται και στόχους για το περιβάλλον και την απασχόληση. Μιλούμε για την περιβαλλοντική αηφορία της γεωργικής πολιτικής και αυτό θα συμβάλλει στους στόχους για το κλίμα και για στη μείωση του ενεργειακού απο... αποτυπώματος, στη μείωση της εξάρτησης από τα ορεικτά καύσιμα και τον άνθρακα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα έχουμε προστιθέμενη αξία. Έχω την αίσθηση ότι ο ρόλος της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορεικτά καύσιμα και τον άνθρακα την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος δηλαδή δεν ε, έχει αξιολογηθεί επαρκώς. Είναι σημαντικό οι πλούσιες χώρες μέλη να συμβάλλουν περισσότερο για να επιτευχθούν οι στόχοι ε, συνοχής από ό,τι το πράττουν τώρα, σήμερα. Δεύτερον, έχω επίσης να πω, ε, συγγνώμη μισό λεπτό, το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να στρέφεται περισσότερο προς τις φτωχότερες χώρες μέλη και να έχει στόχους κλιματικούς και στόχους απασχόλησης μιλούμε εκεί και για εκπαιδευτικά προγράμματα. Να συγκεντρωθούν τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής στις πιο φτωχές χώρες και αυτό θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική σύγκληση και θα ε, κομίσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, καθώς το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ωφεληθεί από την οικονομική σταθερότητα στις χώρες συνοχής. Ταυτόχρονος είναι απαραίτητο να ενισχυθεί περισσότερο η διοικητική ικανότητα των ε, ε, πιο φτωχών ε, αποδεκτριών χωρών. Και αυτό έχει τονιστεί στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτον, οι δαπάνε ερευνητικέ για την έρευνα και την κοινοτομία θα πρέπει να αυξηθούν με έμφαση ιδιαίτερη σε πτυχές που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και το περιβάλλον. Δεν μιλούμε μόνο για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο, αλλά και τις επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην εκπαίδευση, να στηρίξουμε την κινητικότητα μαθητών, φοιτητών και νεαρών ενηλίκων γενικότερα. Τέταρτο, δαπάνες για διασυνοριακές υποδομές στραμμένες προς την αηφορία. Μιλούμε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, για το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη, Interconnecting Europe, και στρατηγική για τη μείωση της ε, ε, ε, ενεργειακής εξάρτησης, για λιγότερες εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και μείωση του κόστους και στις υδροδρομικές και άλλες μεταφορές. Καθαρή ενέργεια, δίκτυα καθαρής ενέργειας. Θα πρέπει η στρατηγική Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, να αξιοποιηθεί ρητά και να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής για τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα. Τέλος, πρέπει να έχουμε συντονισμένη προσέγγιση για το μετριασμό των επιπτώσεων από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Αυτό ορίστηκε στη Σύνοδο σχετική και στις 16 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άρα περιλαμβάνονται περισσότερα κονδύλια για τη βοήθεια, για την αποτροπή, για τα προγράμματα μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, για την υλοποίηση πολιτικών ε, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης. Και τέλος, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να ε, ε, υιοθετήσει τους επίσημους στόχους για την ανάπτυξη αναπτυξιακής βοήθειας και να τους στηρίσει και να γίνουν τα δέοντα. Οι δαπάνες για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να λάβουν χώρα στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να αυξηθούν οι στόχοι, να αυξηθεί ο πύχης από το 20% να ενισχυθεί και να αυξηθεί ο στόχος που έχει να κάνει με το πόσο συμβάλλει η πολιτική γεωργία στην κλιματική πολιτική στην πολιτική για το κλίμα. Όλα αυτά θα φέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο στόχος της αηφορίας να επιδιωχθεί ανεξαρτήτως του ποιο από τα πέντε σενάρια θα ακολουθηθεί τελικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματο είναι ο στόχος για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. και είναι αρκετό για να έχουμε αλλαγές και νέες προτεραιότητες στον κοινοτικό προπολογισμό. Ακόμα και αν κάνουμε αλλαγές, τι αλλαγέ που θέλουμε, τις πολύ μεγάλες και στον τομέα τη γεωργία και στον τομέα τη συνοχή. Δηλαδή, οι περικοπές στις ε, γεωργικές ενισχύσεις, θα μας επιτρέψουν να έχουμε αυξημένες δαπάνες σε έρευνα, σε καινοτομία, σε περισσότερη εφορία και θα δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό σε κάθε τομέα δαπανών και όλα αυτά θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών δαπανών κυρίως σε τομείς που χρειάζονται περισσότερη ενοποίηση και ολοκλήρωση και αν η ομάδα κρατών μελών εμπλέκεται περισσότερο και ενδιαφέρεται περισσότερο, τότε αυτό σημαίνει ότι θα βαθύνει η συνεργασία αυτών των χωρών και άρα η ενοποίηση και ολοκληρωσή τους. Integration. Και για να φανούν αυτές οι δομικές μεταστροφές, οι αλλαγές και οι προτεραιότητες, θα πρέπει να προσαρμοστεί ο βασικός τομέας βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε και διάφορες επικεφαλίδες, άλλους τίτλους, ε, ε, καινοτομία, εκπαίδευση, υποδομές με χαμηλή, χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, άλλους ε, υποτομέας και τομέας να είναι η μετανάστευση, αναπτυξιακή βοήθεια, εσωτερική ασφάλεια ασφάλεια των συνόρων, άμυνα και διοίκηση. Να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου εδώ με κάποια σύντομα συμπεράσματα και μια σύντομη επισκόπηση. Σε γενικές γραμμές, κλειδί, στοιχείο κλειδί για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για το 2020 είναι η περιεκτική και αηφόρος στρατηγική. Θα αυξηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που δημιουργούν οι δαπάνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναθεωρηθούν, μεταρρυθμιστούν θεμελιωδώς οι δαπάνες και αυτό είναι απαραίτητο για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το θέμα των ιδίων πόρων, να αδράξουμε το momentum, την ορμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή και πρέπει να προχωρήσουμε με αυτές τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό και αυτό το τόνισε και η ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους, ότι το Brexit δηλαδή είναι μια ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε θέμελα τη διάρθρωση και δομή των ευρωπαϊκών δαπανών αλλά και των εσόδων. Μέσα από διαφορετικούς διάβλους το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα ήταν κατά της προοπτικής της καθαρής θέσης και εστίαζε την προσοχή στη διαφορά μεταξύ των εισφορών στον κοινωνικό προϋπολογισμό και μεταφορών που εισέπρατε από τον προϋπολογισμό. Αυτό καταρχάς και μετά δεν θα χρειαστεί και η έκπτωση, το rebate προς το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Άρα μπορούμε να έχουμε ε, την κατάργηση των διορθωτικών μηχανισμών και τέλος το Brexit μπορεί εμέσως να στηρίξει τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο διότι θα αυξήσει τη γνώση σε επίπεδο κρατών μελών. Θα καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός πρέπει να φέρνει περισσότερο προστιθέμενη αξία. Ε, για να πιστούν και οι πολίτες καλύτερα για την αξία αυτού. Και έτσι ε, η αποδοχή των μεταρρυθμίσεων ε, θα είναι μεγαλύτερη και σε επίπεδο δαπανών και σε επίπεδο εσόδων. και μπορεί και να ενισχυθεί η αποδοχή των πολιτών σε διάφορους φόρους ε, που μπορεί να επιβληθούν, όπως είναι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών και χρηματιστηριακών συναλλαγών, ε, διότι αυτοί θα μετατραβούν σε μέρος των εσόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού. Πρέπει να έχουμε συνολικές λύσεις, σε λύσεις σε πακέτο, σε επίπεδο δαπανών και σε επίπεδο εσόδων. Ένα βασικό παράδειγμα είναι η συγκέντρωση των Ταμείων Συνοχής στις φτωχότερες χώρες μέλη, οι οποίες στην πλειοψηφία τους αυτή τη στιγμή έχουν αντίρρηση στις συντονισμένες προσπάθειες περικοπών, γιατί είναι ένα από τα εργαλεία που έχουν για ανταγωνιστικότητα. Και αυτό θα μπορούσαμε να το δεχθούμε ως αντάλλαγμα ε, του να δεχθούν τη συμφωνία για ίδιους πόρους που θα βασίζονται στη φορολόγηση και μετά μπορούμε να έχουμε ε, επιβαρύνσεις και τέλη στον άνθρακα και στα ορυκτά καύσιμα για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού ε, και αυτό θα είναι κίνητρο για τις ε, χώρες αυτές, για διάφορες χώρες, προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους την ενεργειακή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα απαντήσω με, ενδιαφέρον στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή παρουσίαση αυτή και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στους εισηγητές και στους δύο εισηγητές ή σε έναν από τους δύο αν θέλει να μιλήσει τώρα η κυρία Τωμά και μετά στους ε, εισηγητές για θέματα πόρων. Βλέπω ότι εδώ είναι οι σκιώδες και όλοι οι σχετικοί συνάδελφοι. Η Ιζαμπέλ Τωμά έχει λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και μετα στους εισηγητες για θεματα πορων βλεπω οτι εδω ειναι η Ισραήλ Τωμά έχει λοιπόν το λόγο Σας ευχαριστώ πρόεδρε Σας ευχαριστώ και ολοι οι σχετικοι κυρία για την παρουσίαση αυτή η οποία ήταν πάρα πολύ εκτενής. Να κάνω κάποιες διευκρινήσεις γιατί σε ό,τι αφορά την κατάρτιση της έκθεσης πρωτοβουλίας αυτής ε, προβλέψαμε οι τομεακές ε, επιτροπές να μας δώνουν τα στοιχεία. Ακόμα και αν συζητάμε εδώ συχνά για θέματα πολιτική συνοχή, νομίζω ότι στην Επιτροπή Προπολογισμού θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακριβεί σε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Και το λέω αυτό και ίσω να προκαλώ σε ό,τι αφορά το θέμα τη χρηματοδότηση. Μιλήσατε για πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχετε και συζητάτε σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή και την, ε, πολιτική, την κοινή πολιτική για τη Γεωργία. Δεν ξέρω αν τα θυμάμαι όλα και τα έχω όλα υπόψη μου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον όμως ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παρουσίασή σας και εδώ συμφωνούμε και με τα συμπεράσματα της, Επιτροπής Προϋπολογισμού είναι ότι μας φαίνεται ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν πόροι για τα αναπάντεχα περιστατικά και αυτό που θα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος είναι να γνωρίζουμε με ποια μέσα θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό ακριβώς πιστεύετε ότι καλύτερα θα ήταν να υπάρχει ένα α, ταμείο, ένα μέσο σε κάθε πολιτική ξεχωριστό ή ένα νέο ταμείο εγκάρσιο και πώς θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί και τι είδους ε, ε, μέσα θα έπρεπε να κινητοποιηθούν. Α, ποια είναι η απόψή σας ε, για κάτι άλλο τώρα, για αυτό που θίξατε σε ό,τι αφορά την αγροτική, τη γεωργική πολιτική. Καταναμένω τι λέτε όταν μιλάτε για την ανάγκη για μια βασική στροφή προς την βιώσιμη πολιτική γεωργία. σε ό,τι αφορά και το τρόφιμα. Αυτό θα μας κοστίσει πολύ. Αν ε, συνεχίσουμε όμως ε, να απελευθερώνουμε την ε, πολιτική, την αγροτική, πιστεύω ότι θα μας στοιχήσει αν κάνουμε αυτό που κάνουν και τα άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα η ΙΠΑ, η Κίνα, που επενδύουν υπέρμετρα. Και είναι πολύ μεγαλύτερε οι επενδύσει του από αυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ισχύει και για την πολιτική συνοχή. Ακριβώ το ίδιο. Αν όντω μειώσουμε τι ε, επενδύσεις μας, τις μας στις πιο φτωχέ χώρες, αυτό που ρισκάρουμε είναι οι υπόλοιποι να υποχωρήσουν σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της πολιτικής συνοχής και σε τελική ανάλυση να παραλύσει. Αν αυτή η πολιτική λοιπόν δεν ωφελήσει τους πλέον αδύναμους, μόνο και μόνο επειδή το θέσατε το θέμα αυτό, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βρούμε μία δομή, ένα τρόπο λειτουργίας, ο οποίος θα μας επιτρέψει παράλληλα, όπως είπατε και εσείς, και να υπάρχει προβλεψιμότητα και ορατότητα και μια μεγάλη επισκόπηση της κατάστασης, αλλά και παράλληλα η πολιτική αυτή των αρθρωτικών ταμείων και να ανταποκρινόμαστε και στις ε, κρίσεις που παρουσιάζονται στα πρόβλεπτα αυτά περιστατικά τα οποία ανακύπτουν και τα οποία δεν προβλέπονται προφανώς επαρκώς στο δημοσιονομικό πλαίσιο. και τα οποία επιφέρουν ε, μεγάλες ε, πιέσεις ε, σε προπολογισμού για τις υποδομές, για την έρευνα και για άλλους τομείς. Κυρίως αυτός που ανέφερα. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αποφύγουμε αυτό και τι είδου μέσο θα χρειαζόταν για να το αποφύγουμε αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Όλμπρεχτ. Ναι, αυτό που θέλω να κατανοήσω είναι το εξή. Προτείνεται να αλλάξει η δομή του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, ναι ή όχι. Και επικεντρώνομαι σε όλα τα στοιχεία που αναφέρουν ότι οι βασικέ επικεφαλίδε ε, θα πρέπει να εστιάζονται στι βασικέ προτεραιότητε. Και μιλάτε για το πρώτο κεφάλαιο, για το πρώτο τίτλο. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Που θα συμπεριλάβει όλο το 1α 2α και 2. Αυτό μπαίνει στο πρώτο, στην πρώτη επικεφαλίδα. Βιώσιμη ανάπτυξη. Και ύστερα έχουμε την μετανάστευση και την ε, δίκηση της ιστορικής ασφάλειας. Ίσως κάνω λάθος, αλλά δεν προτείνεται και επαναστατικές αλλαγές, μάλλον τεχνικές προσαρμογές θα έλεγα, στη σημερινή κατάσταση. Σωστά λοιπόν καταλαβαίνω. Δεν πιστεύετε ότι αυτές οι αλλαγές αποτελούν το ουσιαστικό πρόβλημα. Το πρόβλημα πιστεύετε ότι είναι κάπου αλλού, ότι δαπανούμε υπερβολικά πολλά μέσα για έναν σκοπό ο οποίος δεν είναι αρκετά ωφέλιμος σε τελική ανάλυση, σε ό,τι αφορά τη συνοχή, ό,τι αφορά τη γεωργία, το οποίο προφανώς ε, δεν θα το δεχτούν πολύ θετικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό αποτελεί λοιπόν ένα στοιχείο. Σωστά κατανοώ μια αλλαγή φιλοσοφία, μια στροφή θα έλεγα. Και δύο μικρέ παντερήσει τώρα επιτρέψτε μου, είσαι Και αυτό σχετίζεται με την πρόκληση, το στοιχείο τη πρόκληση το οποίο θα ήθελα να συμπεριλάβω. Πρώτον, για μισό λεπτό να βρω τη διατύπωση. Σε ό,τι αφορά την υπερβολική συγκέντρωση. Μα πού είναι. Στην τέταρτη διαφάνεια. Για την τοπική προστιθέμενη αξία. Εξ ε, καταλαβαίνω, το λέτε με αρνητική χρειά αν υπάρχει τοπική προστιθέμενη αξία, δεν είναι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι πολύ αμφιλεγόμενο, γιατί έχουμε τι ευρωπαϊκέ προτεραιότητε. Έχουμε διάφορου τρόπου ε, για να πετύχουμε ακριβώ αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και σε κάποιε περιπτώσει περνάμε από το τοπικό επίπεδο. Α, σε τοπικό επίπεδο μένει ευρωπαϊκή όμω προστιθέμενη αξία και πάλι. Και το δεύτερο στοιχείο είναι οι συμφωνίε πακέτου είναι το ίδιο με την ρεσιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πακέτο, τι σημαίνει. Είτε το δεχόμαστε ολόκληρο, είτε το απορρίπτουμε ολόκληρο, αλλά μιλάμε και για αιρεσιμότητα σε διάφορε πολιτικέ. Το ίδιο λοιπόν εννοείται, ή μήπω υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του στοιχείου αυτού και τη αιρεσιμότητα στι διάφορε πολιτικέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα να περάσουμε στου σκιώτε εισηγητέ. Από το ECR, ο Μπεν Χόλμερ, θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα ιδιαίτερω να ευχαριστήσω για την πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Και χαίρομαι που τώρα μας κάνετε την παρουσίαση αυτή, γιατί αλλιώς θα με κατηγορούσαν οι συνάδελφοι ότι αντιγράφω όλα τα επιχειρήματα τα οποία αναφέρετε, γιατί ξέρετε μου μιλήσατε κατευθείαν μέσα στην καρδιά μου και θα ήθελα να πω δύο πράγματα, γιατί θεωρώ ότι αποτελούν και τα σημεία κλειδί, αν θέλετε. Αυτό που παρατηρούμε στην παρούσα φάση, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι μια δραματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία και πρέπει να ανταποκριθούμε και προφανώς πρέπει να ανταποκριθούμε και από πλευρά στον προπολογισμό. Δεν μπορούμε πια να αγνοούμε το γεγονός αυτό. Και το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι το εξή τι θα κάνουμε. Θα πούμε ότι έχουμε πάρα πολλέ απαιτήσει δικαιολογημένε και μπορούμε να τι πετύχουμε μόνο αν έχουμε πιο πολλά χρήματα και θα πρέπει να κάτσουμε να υπολογίσουμε πόσα χρήματα θέλει και χρειάζεται ο καθένα. Νομίζω ότι αν καταρτήσουμε διάφορα τέτοια σενάρια, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να αποφασίσουμε και πόσο θα κοστίσουν και πώ θα πρέπει να τα πληρώσει τελικά. Κάτι άλλο. Αν ε, κάπου διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν όρια τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν, θα πρέπει να τηρήσουμε αυτά τα ανώτατα όρια και έτσι να αποφασίσουμε ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και κάποια άλλα όχι. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μία μορφή δικαιοσύνη ε, έναντι των πολιτών. Νομίζω ότι είναι απόλυτα εσφαλμένο να διατηνόμαστε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι διανόητο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε. Και έτσι περνάμε στο επόμενο σημείο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θεωρεί ότι είναι υπεύθυνη και αρμόδια. Μιλάμε για την κοινή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και όλοι μιλούν για την ενίσχυση της αρχής της επικουρότητας. Αλλά εγώ πρακτικά καταλαβαίνω κάτι διαφορετικό, να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Πού μπορούμε να πετύχουμε κάτι και πού βρίσκονται τα σημεία προτεραιότητά μα, Για παράδειγμα, στον τομέα τον αγροτικό. Εδώ και κάποιε ημέρε αυτό που ζητώ είναι να θέσουμε νέα σημεία προτεραιότητας και να κάτσουμε να κοιτάξουμε πού θα πρέπει να δράσουμε με γνώμονα το μέλλον. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ε, πολιτική συνοχή. Αν υποστηρίζουμε και ενισχύουμε εδώ και δεκαετίες μία περιφέρεια στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, χωρίς να σημειώνονται ιδιαίτερη πρόοδο, θα πρέπει κάποια στιγμή να ρωτηθούμε αν υπάρχει αποτέλεσμα και αν υπάρχει επιτυχία στην πολιτική μα αυτή. Γιατί αν έχει λειτουργήσει η πολιτική συνοχή, θα πρέπει να έχουν μειωθεί κάπω τα συγκριτικά μειονεκτήματα τη περιοχή αυτή. Ιδάλω, ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε μήπω ε, κάποιε επιδοτήσει έχουν περάσει σε μια φυσιολογική κατάσταση και έτσι εισπράττονται. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε κατά πόσον θα συνεχίσουμε να ξοδεύουμε τα χρήματά μας έτσι, κατά πόσον η δαπάνη αυτή είναι βιώσιμη και ευφυής. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες θα συμπεριληφθούν στη Λευκή Βίβλο ασφαλώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου και θα περιλαμβάνονται διάφορα σενάρια. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσουμε λοιπόν τι θέλουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε και να μην ξεχνάμε πάντα το σκέλος της χρηματοδότησης για να ξέρουμε τι θα κοστίσει και πόσο. Ευχαριστώ. Επόμενος σκιώδης, αν θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Ντεπρέ από τους Φιλελεύθερους. Um, the shadows. Now Πρώτα οι σκιώδεις για αυτή την έκθεση και μετά οι συγγητές για το θέμα των ίδιων πόρων. Πρόεδρε, άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση. Ήταν μια διανοητική άσκηση. Ε, αυτά που μας είπε η εμπειρογνώμονα. έχει πάρα πολλές ιδέες, οι οποίες μπορώ να συμμεριστώ. Όμως φοβάμαι ότι ένα σημαντικό κομμάτι των προσανατολισμών που προτείνεται από την εμπειρογνώμονα ε, είναι σε διαφορά φάσεις με τις ανησυχίε ανησυχίες που θα εκφράσουν διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και δεν εκφράζω αξιολογική κρίση εδώ καθόλου. Αν λάβω υπόψη μας ε, την, ανησυχίε τις ανησυχίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θεωρώ πως αυτό θα γίνει. Και το, αν λάβω υπόψη το συντηρητισμό τους, θεωρώ ότι θα έχουν δυσκολίες να δεχτούν κάποιους από τους προσανατολισμούς που μας πρότεινε η εμπειρογνώμονα. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ 100% με αυτό που εξηγήσατε για τις βασικές αρχές του προπολογισμού μας που θα πρέπει να αλλάξουν και να ευθυγραμμιστούν με, τις νέες, με τους νέους προσανατολισμούς. Δεν νομίζω όμως ότι η συζήτηση με το Συμβούλιο θα αφορά αυτά τα στοιχεία. Θεωρώ ότι το κέντρο βάρος θα δοθεί αλλού, θα είναι αλλού. Παρ' όλα αυτά, ε, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ ακούγοντας και διαβάζοντας δύο πράγματα που είπατε πολύ συγκεκριμένα. Το ένα λέει ότι η ικανότητα να λαμβάνουμε ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να εξαρτάται από τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου. Ότι θα πρέπει να σέβεται κανείς το σύνολο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι μια πολύ βασική αρχή. Επίσης, ε, ε, σοκάρουμε πάρα πολύ που βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάποια κράτη-μέλη τα οποία λαμβάνουν τα περισσότερα κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν έχουν προσυπογράψει σε θέματα όπως παραδείγματο χάρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει σαν σκοπό να καταπολεμήσει την απάτη εναντίον των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα έλεγα όχι ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δεν αναγνωρίζουν την ε, νομιμότητα και το ρόλο και τις αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Ξέρω ότι διάφοροι φίλοι δεν θα δεχτούν αυτή τη λογική, τη δική μου λογική, αλλά έπρεπε να το πω γιατί το θεωρώ απαραίτητο και συνεπές πολιτικός πώς. Δεύτερον, δεύτερο στοιχείο το με το οποίο συμφωνώ. Όταν λέμε ότι τα ταμεία συνοχής θα πρέπει να πάνε περισσότερο σε αυτούς που τους έχουν ε, ανάγκη παρά ε, Προ πλούσια, τα πλούσια κράτη-μέλη. Θα πρέπει να πείσουμε όμω τα κράτη-μέλη τα οποία θεωρούν ότι είναι καθαροί εισφορεί. Ε, ιδεολογικά συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να το συνδυάσουμε με του στόχου προστασία του κλίματο, με του στόχου για την προστασία του περιβάλλοντο και μια πολιτική ε, έτσι, προορατική για την μετανάστευση και την ένταξη των ε, μεταναστών. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που υπόθηκε και νομίζω ότι θα είναι από τα βασικά στοιχεία, αλλά δύσκολα και λεπτά στοιχεία της μελλοντική διαπραγμάτευσης που θα έχουμε. Όταν συζητήσουμε το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Από, τους πράσι, από, του, την ΚΟΕ, Λίαν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή και θα Ήθελα να σχολιάσω το εξή. Ο κοινωνικό πυλώνα νομίζω ότι λείπει από πολλέ ε, πτυχέ τη παρουσίαση. Μιλάμε για την ενεργή των νέων. Πρόκειται για μία δήλωση η οποία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά από του νέου μα και λέμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στου νέου μα, αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια διαφορά, να σημειώνεται κάποια διαφορά. Και ένα λόγια. Ποια είναι λοιπόν η λύση στην πρόκληση αυτή. Αν κάνουμε μία μικρή επένδυση σε κάποιο σκέλος στον κόσμο, στον Horizon, η απόδοση της επένδυσης είναι τεράστια. Αυτή την επιχειρηματολογία νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε, παρά να λέμε διαρκώς ότι θα πρέπει να επενδύσουμε και στην ουσία να μην το κάνουμε ποτέ. Τι και το θέμα της σε πολλές χώρες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλά ήδη επενδύονται στην ΚΑΠΑ και υπάρχει ενδεχομένως πιο αποτελεσματικός τρόπος ε, αντιμετώπισης του θέματος, να κοιτάξουμε την επιστική ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Να μην επαναλάβω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, αλλά να πω το εξή. Θα ήθελα να κοιτάξω πιο λεπτόμερως αυτά τα πακέτα, τις συμφωνίες πακέτο που αναφέρεται και το πώς θα καταφέρουμε με τον τρόπο αυτό να βγάλουμε τον κόσμο από την φτώχεια και οι επενδύσεις σε χαμηλή στη ενέργεια χωρίς άνθρακα και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις κλειδονισμούς αυτούς τα σοκ αυτά και πώς θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα εργοστάσια που κλείνουν τον αντίκτυπο στο εμπόριο θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και πιο μακροπρόθεσμα όσο μπορούμε να προβλέψουμε γιατί ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τι έχετε να πείτε από αυτού. Προσβλέπω σε μια συζήτηση πιο λεπτόμερη και μακροσκελής. Και κλείνοντα, να πω το εξή: Θεωρώ ότι είμαστε τόσο απομακρυσμένοι από τον κόσμο, από του πολίτε. Υπάρχει τόσο απαγοήτευση και αγανάκτηση ε, και παρανόηση σε ό,τι αφορά το τι ακριβώ κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χρηματοδοτεί. Δεν καταλαβαίνουν τι διαδικασίε υποβολή αιτήσεων που δυσκολεύουν τα πράγματα με τον πολίτη που θεωρώ ότι θα πρέπει να το θέσουμε αυτά σε επίπεδο εθνικού διαλόγου. Να αναφέρουμε τα μέλη, για παράδειγμα, ΜΚΟ και το καθεξής. Να τους ενημερώσουμε, να καταλάβουν αυτοί τουλάχιστον τι είναι ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και γιατί πρέπει να ψάχνουν πόρους, να κάνουν αιτήσει κτλ. Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να γίνει αυτή η δικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο πρόεδρος. η πράσινη δεν τους βλέπω στην αίθουσα, το EFTD απόν και το είναι e απόν. Να δώσω το λόγο στο Γιάννη Λαμπαντόφσκι που είναι συγκεκριτή για τους ιδίους πόρους τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι τόσο ειδικό για τους ιδίους πόρους. Ε, επικεντρώνομαι σε πρακτικά χρηματοδοτικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά δηλαδή εμπειρογνωμοσύνη επί της πράξης και ασχολούμαι πιο πολύ με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τις επενδύσεις. Αλλά το θέμα αυτό ασφαλώς αφορά και την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τον πολίτη, σε ό,τι ρόλο στη Σαξονία. Η Ευρώπη γίνεται ορατή και προβάλλεται μέσω της νομοθεσίας και αυτό δεν αρέσει πάντα στους πολίτες μας και μάλιστα συχνά τους προκαλεί δυσαρέσκεια αλλά και μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος, του ευρωπαϊκού οράματος εδώ είναι πιο θετική η επίδραση. Το παράδοξο λοιπόν, κυρία Σάτσιν Στάλερ, είναι το εξή, ότι όσο πιο περιφερειακό είναι το πρόγραμμα, τόσο πιο πολύ προβάλλεται και τόσο πιο πολύ προβάλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θεωρείται ότι είναι άχρηστο κομμάτι του προπολογισμού, αλλά όσο πιο πολύ προστιθέμενη αξία έχει το πρόγραμμα αυτό, και εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Υποστηρίζω απόλυτα τέτοια προγράμματα. Όσο πιο ευρωπαϊκό είναι, τόσο πιο απόμακρο και λιγότερο προβεβλημένο είναι για τους ε, πολίτες. Και έτσι δεν το προσπίζονται, δεν το υποστηρίζουν. Αυτή είναι η πρακτική, αν θέλετε, πλευρά των δημοσιονομικών προοπτικών μέχρι το 2020 σε διαφορά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ο ορίζοντας ε, αυξήθηκε Connecting Europe 150% 50% ταμείο ανάπτυξη και αυτό που μειώθηκε ήταν η συνοχή και η γεωργία. Αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το εξή ε, ως μάθημα από το τι συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αρχικά το πρόγραμμα, το project, το έργο αυτό. Τι, πού ήταν οι περικοπές ε, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις τέτοιων έργων. Μιλήσατε για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για μέλλοντο τραφή πολιτική. Πολλοί μιλούν για μάλλον ε, περικοπές στον ορίζοντα, στην ασφάλεια. Και αυτό το οποίο προσπιστήκαμε πιο στεναρά ήταν η κοινή αγροτική πολιτική με μοναδική εξαίρεση την Σουηδία, η οποία δεν ε, υποστηρίζει ιδιαίτερο στην ΚΑΠ παρά τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα αυτό. Πέρα από το να σκεφτόμαστε το μέλλον, η πρακτική ανάλυση του τι ήδη έχει συμβεί στις διαπραγματεύσει θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη των μελλοντικών πολιτών, πολιτών συνομικών προοπτικών. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο Ζεράρα, ε, θα πρέπει να παταχθεί η διαφθορά και να συνδέονται οι πόροι το... μάλλον δεν συμφωνώ το να συνδέεται η χρηματοδότηση με κάποιου όρου, γιατί ουσιαστικά κυβερνείται, τιμωρείται ο λαό για λάθη τη κυβέρνηση, τη δίκηση. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να προσέλθω. Σας ευχαριστώ κύριε Μιρεσάν που προεδρέσατε στη θέση μου. Φαντάζομαι ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αρχική σας συζήτηση. Ήμουν στην Επιτροπή Γεωργίας. Δεν έχει κανένα νόημα ε, να, φτάνουμε τους, να φέρνουμε στο, στο σημείο της στόχευσης τους γεωργούς λόγω των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου που συνάπτουμε. Λοιπόν, Κλείνω αυτήν την παρένθεση. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Ε, ορισμένοι βλέπετε το Brexit ως ε, ευκαιρία. Οι περισσότεροι από εμά το, το βλέπουμε όμως ως καταστροφή και για τους μεν ναι και για τους δε. Στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης χθε ε, συμφωνήσαμε σε μια γνωμοδότηση που υπερψήφισαν 27, κρατη, 27 βουλευτές υπέρ, 4 ε, την καταψήφισαν. Ε, μιλάω για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην Επιτροπή Ρέτζι υπάρχει ανησυχία για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ξέρουμε ότι στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν, ίσως και στο Κοινοβούλιο, η πολιτική συνοχή δεν έχει πολλούς οπαδούς. Φοβόμαστε ότι απειλείται στο μέλλον η πολιτική αυτή. Εάν υπάρχει μια περικοπή στον προπολογισμό λόγω Brexit, φοβάμαι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των περικοπών ε, θα το υποστεί η περιφερειακή ανάπτυξη. Το φοβάται αυτό η Επιτροπή Ρέτζη και θα ήταν λάθο. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του Πουδουπού, για πρώτη φορά η Επιτροπή μου λέει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το 5 5 Αλλάξαμε τη θέση μας δηλαδή εδώ. Όπως είπαν και άλλοι όμως θα θέλαμε μια σοβαρή αναθεώρηση μετά από πέντε χρόνια. Ξέρουμε ότι σήμερα στο Πουδουπού κάνουμε τη διάμεση αναθεώρηση στα μέσα, αλλά είναι μια τυπική διαδικασία. Θα πρέπει να έχουμε το 5 συν 5 χρόνια και στα 5 χρόνια να κάνουμε μια σοβαρή αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και να θεωρήσουμε και τα προγράμματα. Επίσης, όλες οι περιφέρειες θα πρέπει στο μέλλον να λαμβάνουν ε, κονδύλια από την πολιτική συνοχής. Ε, διαφωνούμε με αυτά που είπατε, ότι μόνο λέει, δηλαδή, τα φτωχότερα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κονδύλια από την ε, πολιτική συνοχής, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και στα πλούσια ε, κρατημέλη. Ακόμα και στα, στις πλούσιες ε, περιφέρειες υπάρχουν και στόχες. Όλες οι περιοχές θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Επιπλέον η πολιτική συνοχής δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση, είναι και πολιτικό κομμάτι. Υπάρχει πολιτικός ε, άξονας. Οι περισσότεροι που ζουν στις περιφερειές μας το μόνο που ξέρουν από τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή η μπλε σημαία και όταν βλέπουν ας πούμε ότι ένα έργο ή ένα project χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν θα πρέπει να προσυπογράψουμε στο επιχείρημα ότι τα φτωχότερα κρατημέλη μόνο θα πρέπει να παίρνουν χρηματοδότηση. Όχι, όλες οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίρνουν κονδύλια. Επίσης πιστεύουμε ότι στο μέλλον η πολιτική συνοχή θα πρέπει να παραμείνει ε, να βασίζεται στις επιχειρήσεις. μικρές οργανώσεις, φυσικά θα υπάρξουν και δάνεια, γιατί ε, όμως ε, οι επιχορηγήσει θα πρέπει να είναι ένα κομμάτι μεγάλο της πολιτικής συνοχής. Αυτά να παίρνουν οι δικαιούχοι. Ε, γιατί υπάρχουν οργανώσεις που θα μπορούν να αποπληρώνουν με δάνεια, μικρές οργανώσεις κυρίω. Επίσης, υπάρχουν πολλά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται για έργα στα πλαίσια των υποδομών, έργα υποδομών. Εγώ θα έλεγα μία είναι η απάντηση. Μεγαλύτερη ευελιξία. Γιατί όλα τα κράτη-μέλη ε, και όλε τι περιφέρειες έχουν διαφορετικέ ανάγκε. Κάποια φτωχά κράτη-μέλη χρειάζονται μεγάλα έργα υποδομών. Ενώ τα πλούσια κράτη-μέλη μπορεί να χρειάζονται λιγότερε επενδύσει στι υποδομέ. Α αφήσουμε λοιπόν μια κάποια ευελιξία εκεί, ούτω ώστε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη και στι περιφέρειε να αποφασίσουν πού είναι οι προτεραιότητέ του. Θα μπορούσαν σε κάποια κράτη-μέλη να είναι περισσότερε υποδομέ, αλλού περισσότερη ανάπτυξη, αλλού περισσότερη κατάρτιση, α πούμε. Αν θέλουμε να εστιάζουμε, επίσης θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο στην απλούστευση. Και εμείς και εσείς είπατε, Πρόεδρε, ότι υπάρχουν ε, πολλά γραφειοκρατικά κολλήματα. Έχουν γίνει προσπάθειες για να έχουμε απλουστευμένες επιλογές. Αυτό που προτείνουμε στην Επιτροπή Ρέτζι είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου ταμείου, ίσως ορισμένοι το θεωρήσουν υπερβολικό, αλλά τουλάχιστον να δημιουργήσουμε μία κοινή δέσμη κανόνων που να διέπουν όλα τα μεγάλα ταμεία. Θα απλουστεύσει πάρα πολύ τα πράγματα για τους δικαιούχους. Και το τελευταίο, πραγματικά τελευταίο, Υπάρχει γενικά συνένεση. Το μόνο προβληματικό σημείο στην Επιτροπή μας αφορά το θέμα το, των μακροοικονομικών προϋποθέσεων και της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Ε, εκεί υπάρχει, είναι η μοίρα του, της έρηδος αυτή. Το μοίρα της έρηδος, συγγνώμη. Είναι τεράστιο θέμα αυτό και πολλοί βουλευτές είναι πολύ δυσαρεστημένοι με την πρόταση αυτή. Όλοι κατάλαβαν ότι πήρατε το λόγο γιατί είσαστε μέλος της Επιτροπής Ρέτζι και ότι εκφράζετε την άποψη της Επιτροπής αυτής. Και τώρα θα ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής ΔΕΒ, της Επιτροπής Ανάπτυξης δηλαδή. Ο κύριος Ρεμπίχ. και αν θα μπορούσατε να περιοριστείτε στα δύο λεπτά γιατί έχουμε καθυστέρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά αυτή τη φορά δεν την πληρώσει, κυρία Τωμά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Πολιτικής, ε, στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, μιλάμε για τους ε, βιώσιμού στόχους της χιλιετίας και νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να δραματίσει κάποιο ρόλο σε ό,τι αφορά τα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το είπε και η ομιλήτρια ότι δεν μπορούμε ασφαλώς να βάλουμε και τις 17 στόχους στο επίκεντρο, αλλά μήπως μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση win-win, αμοιβαία επωφελή για την Ευρώπη, όπου έχουμε 20% παραγωγή σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ μέχρι το 2020, μπορούμε να σκεφτούμε μήπως μπορούμε στο στόχο αυτό να βάλουμε το 30% της παραγωγής, γιατί σε τελική ανάλυση η ευημαρία επιτυγχάνεται μόνο εφόσον κάτι παράγεται. Ξέρω ότι η αριστερή πτέρυγα είναι πολύ καλή στην κατανάλωση του κοινοβουλίου. Αλλά και σε διάφορα θέματα δικαιοσύνη. Αλλά νομίζω ότι για να υπάρχει κάποια ισορροπία, ε, σημαντικό είναι να παράγουμε κιόλα. Δεν μπορούμε να παράγουμε μόνο με μικρομεσαίε επιχειρήσει, Εδώ φυσικά αυτό έχει μπει ω προτεραιότητα, αλλά και στην Ήπετρο. Άρα, ποιοι είναι οι στόχοι, οι βιώσιμοι στόχοι της χιλιετίας θα πρέπει να αναπτυχθούν στην Ήπετρο για να δημιουργηθεί και εκεί η ευημερία. Δύο είναι οι στόχοι που θα πρέπει να μπουν ε, στο επίκεντρο. Ο στόχος 6 και ο στόχος 7. Νερό και υγειονομικές ε, εγκαταστάσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες και νόσοι που ακριβώς σε αυτό οφείλονται. Και για να τα πετύχουμε όλα αυτά χρειάζεται ενέργεια, γιατί χωρίς ενέργεια δεν γίνεται τίποτα. Ανανεώσιμες λοιπόν ε, πηγές ενέργειας στην Ήπεθρο και φυσικά με την αντίστοιχη κατάρτιση θα πρέπει όλα αυτά να εγκατασταθούν, να πολιθούν, να υπάρχουν προγράμματα μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ των οικογενειακών επιχειρήσεων σε αυτούς τους στόχους, σε αυτές τις περιοχές ανάπτυξης. Και εδώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει μια νέα προσέγγιση που να είναι ενδιαφέρουσα και για όλες τις πλευρές και να επιτρέψει και την κατανάλωση σε τελική ανάλυση. Αν επιτρέψουμε λοιπόν την κατανάλωση και αν η θέση απασχόληση, αν η εργασία δεν προλογείται τόσο πολύ στο σήμερα, θα υπάρχει και πιο πολύ ισότητα και δικαιοσύνη. Όσο πιο πολύ παράγεται, παραγωγή υπάρχει, τόσο πιο, πολύ εύκολα, τόσο πιο εύκολα θα πετύχουμε το στόχο του ποσοστού ΑΝΑΕΠ για την καταπολέμηση και τη φτώχεια. Για τη συντελική ανάλυση, η φτώχεια μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με κατάρτιση, με υποδομές, με έρευνα για αγαθά υπηρεσίες και φορολογία των όσων, ε, όσο χαμηλότερα γίνεται φορολογία των εργαζομένων. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντική προσέγγιση για την Ευρώπη. Θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να δώσουμε και κίνητρα, κίνητρα προκειμένου οι χαμηλότερες μισθολογικές τάξεις, οι οποίες ε, είναι σε μειονεκτική θέση στην Ευρώπη, γιατί του καταργούνται πάρα πολλά πλέον Θεωρώ λοιπόν ότι αυτέ οι χαμηλότερε μισθολογικέ τάξεις θα πρέπει να υποφελούνται από την εργασία του και να μην υπάρχει μεγάλη ανακύκλωση στο μίσο που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πολλή δουλειά. Και όλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο σημαντικό και στο πολιτικό-μεσονομικό πλαίσιο. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ο κ. Φερνάντε. Κάποιε ερωτήσει, επιτρέψτε μου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους ε, υπεύθυνου τη έρευνας αυτή για τις ε, εμπειρίες που μοιράστηκαν μαζί μας. Καταρχά λοιπόν τώρα να πω το προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι που αναφέρονται στην έρευνα προκειμένου να υποστηριχθεί η ατζέντα της Ευρώπης 2020, η βιώσιμη ανάπτυξη και η συμφωνία του Παρισιού. Το πρώτο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι τι είδους προπολογισμού θέλουμε. Αν δεν εξετάσουμε, δεν αρκεί να λέμε ότι δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Το θέμα είναι γιατί δεν τους πετυχαίνουμε τους στόχους και τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Άρα, γιατί ποσό μιλάμε, τι ποσό χρηματοδότησης ε, μιλάμε, γιατί έχω την αίσθηση εδώ στο έγγραφο αυτό ότι θεωρείται ότι θα συνεχίσουμε με τα ίδια ποσά σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το βασικό ποσό, το βασικό θέμα είναι το επίπεδο χρηματοδότησης το οποίο επιθυμούμε για το πολιτισμό κοινωνικό πλαίσιο. Αν υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το πώς ορίζεται η προστιθέμενη αξία. Τι αποτελεί η προστιθέμενη αξία. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αν μας ε, βοηθούσε να καταλήξουμε σε έναν ορισμό της προστιθέμενης αξίας. γιατί υπονοείται ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία όταν υπάρχει υπερεθνικός χαρακτήρας. Αλλά ουσιαστικά αυτό επιτρέπει τη συνέχιση των περιφερειακών διαφορών. Αν ε, δεν υποστηρίξουμε ότι η προστιθέμενη αξία είναι μόνο τοπική, αυτό αποτελεί ε, από μόνο του αντίφαση. Ύστερα κάτι άλλο. Υπονοείται ότι η πολιτική συνοχή είναι μόνο για τις χώρες των ταμείων συνοχής. Άρα εξαιρείται τις ε, περιφέρειες που είναι φτωχέ σε πλούσιες χώρες, αν καταλαβαίνω σωστά. Άρα το ερώτημά μου είναι ότι η πολιτική συνοχή δεν πρέπει να προορίζεται για όλες τις χώρες, μόνο για κάποιες χώρες, μόνο για κάποια κράτη-μέλη. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν ε, την πολιτική συνοχή ακόμα και οι χώρες που δεν ε, αποτελούν τέτοιες περιοχές. Τέλος, σε ό,τι αφορά την τήρηση τη υφιστάμενη νομοθεσία. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν το υφιστάμενο δίκαιο. Μπορούν, για παράδειγμα, να θέσουν θετικά κίνητρα. Όποιο πληρεί του όρους έχει δικαίωμα για πιο πολύ χρηματοδότηση. Αυτό είναι το σημείο κίνησης και πιστεύω ότι δεν μπορούν να τιμωρούνται οι δικαιούχοι σε περίπτωση σφάλματος της δίκησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ε, μόνο αντιευρωπαϊκά συναισθήματα μπορούμε να προκαλέσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να τιμωρούμε τις επιχειρήσεις, τους φοιτητέ. Αν δεν συμπεριφέρεται σωστά η κυβέρνηση μιας περιφέρειας. Αν κάποιον θέλουμε λοιπόν να τιμωρήσουμε, να τιμωρήσουμε τις περιφέρειες. κυρία Γκαρθία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω ε, με μεγάλη συντομία. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή για το πώς πρέπει να είναι το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συμφωνώ με ορισμένους ορισμούς και με ορισμένες αναλύσεις της κατάστασης, αλλά όχι με τις λύσεις που προτείνεται. Σημερίζομαι τις προκλήσεις. Όντως, αυτό είναι οι προκλήσεις. Οι ανισότητες οι η κλιματική αλλαγή, οι πρόσφυγες, η αύξηση του κινδύνου για φτώχεια. Συμφωνούμε με όλα αυτά, αλλά η λύση στα προβλήματα αυτά δεν είναι η αλλαγή της δομής και διάρθρωσης του ΠΔΠ. Η δομή του ΠΔΠ μας χρησιμεύει για να εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μας χρησιμεύει για να αφηγηθούμε την ιστορία των πολιτικών. Αλλάζοντας τη δομή και τη διάρθρωση δεν θα λύσουμε τα προβλήματα και μακάρι να ήταν και τόσο απλό όσο αυτό που προτείνεται. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να έχουμε αρκετά ανοιχτό ορισμό της προστιθέμενης αξίας. Πράγματι, οι ευρωπαϊκές δράσεις έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ότι οι δράσεις που θα είχαν μόνο εθνικό χαρακτήρα. Στις υπόλοιπες διαφάνειες ασκείται πολύ ισχυρή κριτική στην κοινή γεωργική πολιτική, στα χρήματα που δίδονται στην κοινή γεωργική πολιτική και εγώ νομίζω ότι αν μια πολιτική έχει αποδείξει την προσθέμενη της αξία ευρωπαϊκά, αυτή είναι η κοινή γεωργική πολιτική, είναι και η μόνη πολιτική που είναι αυστηρά ευρωπαϊκή. Κανείς δεν αφισβητεί ότι πρέπει να αλλάξει και να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση η προστιθέμενη αξία της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι κάτι που πολύ εύκολα μπορούμε να υπερασπιστούμε και τουλάχιστον σε οικονομικούς όρους. Για τα, τα λοιπά δεν θα μπω σε σχόλια. Συμφωνώ πολύ με την κυρία Μπόκ ε, με τη θέση της Επιτροπής ε, για τις Περιφέρειες. Είπαμε ότι πρέπει να αυξηθεί το κονδύλι για την εκπαίδευση, για την έρευνα, για την καινοτομία, για τις διασυνοριακές, αν θέλετε, υποδομές. Το, με όλα αυτά συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε από πού πρέπει να πάρουμε τα χρήματα, γιατί δεν θέλουμε να μειωθούν ούτε τα χρήματα της κοινή γεωργικής πολιτικής, ούτε τα κονδύλια της κοινή περιφερειακής πολιτικής. Ένα ερώτημα. Λέτε ότι υπάρχουν πολλά project ή έργα που χρηματοδοτούν και έχουν τοπική μόνο προστιθέμενη αξία. Τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους εγγυγραμμένους στον κατάλογο των ομιλητών. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω δύο σχόλια επιπροσωπικού. Η κοινή γεωργική πολιτική στοχεύει στο να διασφαλίσει ένα συγκεκριμένο εισόδημα για τους γεωργούς. Λέτε ότι τα κονδύλια της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν παρουσιάζουν συνοχή με την συμφωνία για τις ελεύθερες συναλλαγές και για το ελεύθερο εμπόριο. Κάποιες πρακτικές όμως του ελευθέρου εμπορίου οδηγούν στη χρεοκοπία ορισμένους οικονομικούς φορείς και καλό θα είναι να αποκτήσουμε συνοχή στην πολιτική μας και συνέπεια. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, όταν δεσμεύονται, δεν δεσμεύονται μέχρι τέλου και οι πληρωμέ ε, με το εμπάροδο των ετών βαίνουν μειούμενε. Επομένω, θέτω το ερώτημα στην εμπειρογνώμονα και στην Επιτροπή. Ορισμένοι και ορισμένε πολιτικέ, ε, συμβαίνει αυτό για ορισμένε. Ε, πάρα πολλέ πολιτικέ χρησιμεύσαν για το τσιμέντο και την πίσα. Για έργα δηλαδή υποδομών. Δεν πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια για την ε, ε, εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων. Έχουμε πολύ, μεγάλες, ε, πολύ μεγάλη ανεργία των νέων. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχή, το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, τέτοιου είδου κονδύλια για να ενθαρρύνουμε τι πολιτικέ επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία, απόκτηση ικανοτήτων προσόντων, ότι είναι εξαιρετικό εργαλείο να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων και να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. των λεχθέντων. Στρέφουμε προς ε, την κυρία Μαγκρίτε Στράτσεν Στάλερ για να απαντήσει και μετά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερος για όλα αυτά Δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα, σαφέστατα. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα, βέβαια μόνο, δεν είναι δικό μου λάθος. Δείχνει αυτό πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση μου είπατε να είμαι εξαιρετικά σύντομη και γι' αυτό θα παρουσιάσω δύο-τρία σχόλια που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά, όλα αυτά που με ρωτήσατε είναι πολύ σημαντικά. Θα τα, τα έχω σημειώσει, θα τα σκεφτώ και στο σπίτι μου, θα επανέλθω και άλλη μέρα, αλλά ε, τώρα θα περιοριστώ σε δύο-τρία σχόλια μόνο. Ως προς τη δομή και τη διάρθρωση του προϋπολογισμού, με ρωτήσατε κατά πόσο θέλω να αλλάξω αυτό ή αν είναι κάτι ε, που είναι μια επαναστατική πρόταση ή όχι, εν Να σας πω ότι οι κατηγορίες ε, των δαπανών είναι σαφείς και μια χαρά. Δεν χρειάζεται να αλλάξουν, απλά πρέπει να αλλάξουν. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι σαν τίτλο, σαν τομέα. Δεν χρειάζονται επιπρόσθετοι τομεί και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περικοπεί κάτι ούτε να διαγραφεί κάτι τελείω. Απλά πρέπει να αλλάξουν μέρο τα κονδύλια από το τάδε τίτλο να πάνε στον άλλον, από το τάδε τομέα να πάμε στον άλλον, είτε και εντό τομέων. Να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερο προσανατολισμό προς την αηφορία. Αυτό καταρχάς. Και δεύτερον, τι εννοώ τα package deals, με τις συνολικές συμφωνίες. Δεν εννοώ την αιρεσιμότητα προαπαιτούμενα conditionality, αλλά να συνδυάζουμε διάφορα item για τα οποία υπάρχουν διάφορα ωφέλη, να μην αντιμετωπίσουμε το κάθε item ξεχωριστά. Διάφορα μαζί για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ κρατών μελών ή ομάδων κρατών μελών. Το carbon levy, ας πούμε, ε, εισφορές τέλη για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, ρηκτά καύσιμα κτλ. Ε, υπάρχει ομάδα χωρών που το θέλει πάρα πολύ. Άλλη ομάδα χωρών ναι, ε, τη είναι πάρα πολύ δύσκολο για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Άρα, αν βάλει κανείς carbon levy αυτά τα τέλη και επιβαρύσεις, μπορεί να τα συνδέσει με αυξημένη ενίσχυση για προγράμματα μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος στην ίδια χώρα. Και κάτι που είναι κάτι σημαντικό πολιτικά. Δεν θέλω να με παρενοήσετε. Νομίζω ότι το σοκ του Brexit είναι πραγματικά καταστροφικό. Αλλά ίσως τούτων λεχθέντων ας βγει και κάτι καλό από αυτό. Ίσως μπορεί να ε, χρησιμεύσει για να καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι κάτι πρέπει να αλλάξουν εν πάση περιπτώσει και ο ε, ε, κοινοτικός προϋπολογισμός μπορεί κάποιο καλό να κάνει. Δεν είμαι υπέρ του Brexit βεβαίως. Και τέλος, πόσα χρήματα χρειάζεστε, με ρωτήσατε. Περισσότερα από ό,τι έχετε τώρα, απαντώ. Όμω δεν θα τα δεχτούν. Πολιτικά δεν πρόκειται να τα περάσετε αυτό, ούτε θα, θα, γίνει με την υφιστάμενη δομή. Άρα από πριν αλλάξτε το σύστημα των ιδίων πόρων. Για να αλλάξετε το σύστημα των ίδιων πόρων πρέπει να αλλάξετε την υφιστάμενη δομή και διάρθρωση μεταξύ δαπανών και εσόδων, αλλά και εντό των δαπανών και εντό των εσόδων. Πρώτα να αλλάξετε αυτά και μετά να συζητήσετε συνολικά για το ύψο το συνολικό όγκο, αν θέλετε, το συνολικό μέγεθο του κοινοτικού προπολογισμού. Ευχαριστώ. Um, thank you, Chairman. Επόμενος ομιλητής, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Καταρχάς να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό, για την ε, μελέτη αυτή και για τα σχόλια, για την προπαρασκευαστική αυτή δουλειά της Επιτροπής, η οποία δουλειά είναι πολύ εντατική έτσι ώστε η Επιτροπή να κάνει τις καλύτερες δυνατές προτάσεις μέχρι από, ε, μέχρι την επόμενη χρονιά. Δεν μπορώ να σας δώσω ουσιαστική αντίδραση από την Επιτροπή, η οποία έχει συζητήσει αυτά τα θέματα επισήμως. Ωστόσο, θέλω κάτι να σημειωθεί και νομίζω ότι και εσείς το παρατηρήσατε. Ότι δηλαδή ο, ο Επίτροπος Έτιγκερ στην πρόσφατη του ομιλία, για παράδειγμα, στη διάσκεψη για το μέλλον των Ευρωπαϊκών ε, Οικονομικών στις 23 Σεπτεμβρίου μίλησε και εκείνος για την έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Για εκείνο λοιπόν αυτή, αυτό είναι το σημείο κίνησης και έτσι θα αναλύσουμε από εκεί και πέρα τις προτεραιότητες και το πού θα δώσει έμφαση στο μέλλον ο κοινοτικό προπολογισμό. Και τα παραδείγματα που ανέφερε ε, στην ομιλία του ήταν τα μεγάλα επιστημονικά έργα, την άμυνα, την προστασία των υδάτων πόρων, τις διασυνοριακές υποδομές και όλα αυτά συνάδουν και συμφωνούν με την παρουσίαση της δόκτωρος Σράτσενστάλερ και σε σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο τα συμπεράσματα του Επιτρόπου Έτιγκερ είναι πολύ πιο ήπια διότι αναγνωρίζει ότι και οι δύο πυλώνες έχουν αποδείξει ε, την αξία τους και η κοινή γεωργική πολιτική και το Ταμείο Συνοχής. Δεν το τραβάει δηλαδή τόσο πολύ όσο η κυρία ε, Σράτσεν Κάποια θέματα συνεχίζουν να μας ταλανίζουν. Ο Επίτροπος Έτιγκερ λέει ότι Πρέπει να υπάρχει μια δομική ισορροπία μεταξύ του να ζητούμε περισσότερες συνεισφορές από τα κράτη-μέλη, εκεί έχουμε το ισχυρό επιχείρημα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και από την άλλη βάζουμε κάποια χαρτιά πάνω στο τραπέζι ε, για να έχουμε ε, ε, και κάποιες περικοπές ουσιαστικά για να έχουμε μια έξυπνη αντιμετώπιση οι μεγάλοι δομικοί πυλώνες δαπανών, π.χ. συνοχή ή π.χ. κοινή γεωργική πολιτική, θα αποτελέσουν μέρος αυτής της ανάλυσης. Αυτό είναι αυτονόητο. Η δόκτωρ Σράτσεν Στάλερ δοκτωρ σράτσενστάλερ ειπε οι άμεσες πληρωμές να μπουν στην κοινή γεωργική πολιτική και σε να υπάρξει και μια προοπτική σε σχέση με τα της συνοχής. Δηλαδή άμεσες πληρωμές και ενισχύσεις μόνο στις φτωχότερες χώρες μέλη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα μια κλαδική και τομεακή πολιτική να συνδυαστεί με στόχο συνοχής. Σε κάθε περίπτωση όντως η κοινή γεωργική πολιτική ίσως θα πρέπει να εστιαστεί μόνο στους φτωχότερους γεωργούς και στις, ε, φτωχε, φτωχές εκμεταλλεύσεις. Να υπάρχει έννοια του κάπιν, δηλαδή κάποια συγκεκριμένη ανώτατη οροφή ενδεχομένως. Αυτό ίσως έχει κάποιο νόημα, αλλά η συζήτηση είναι στο μέσον της. Και και προσωπικά έχω ένα σχόλιο να κάνω, προσωπικό σχόλιο να σας πω ότι η μεγαλύτερη υπέρμαχη των μεγάλων ποσών και των μεγάλων κονδυλίων της κοινή γεωργικής πολιτικής φεύγουν. Και οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι και οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις των ενισχύσεων αποχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως εκεί μη παραμείνει κάποιος χώρος μετά από το Brexit. Τώρα, ως προς τους ίδιους πόρους, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά θέλω να σας εφιστήσω την προσοχή ε, στο εξή ζήτημα που αναφέρατε και εσείς για μια δημοσιονομικά ουδέτερη προσέγγιση και αυτό είναι σημαντικό για τη συζήτηση των, της χρηματοδότησης στο μέλλον. Δηλαδή, η χρηματοδότηση στο μέλλον θα είναι ε, δημοσιονομικώς ουδέτερη, δεν θα υπάρχει έξτρα επιβάρυνση φορολογική στο φορολογούμενο. Αυτή είναι προσέγγιση βασική στην ομάδα Monte, Monte Group Conclusion, είναι βασικό στα συμπεράσματα αυτά. Άρα εκεί δεν μπορούμε να προβάλλουμε το επιχείρημα ότι ένα νέοι ήδη πόροι θα διευκολύνουν στο να κλείσουμε το κενό που θα δημιουργηθεί λόγω Brexit. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κόψουμε τόσο πολύ γιατί θα υπάρξει Brexit, άρα δεν θα πάρουν χρήματα τόσο πολλά ή μιλούμε για ψηλότερε δαπάνε, άρα για υψηλότερο φορολογικό βάρος. Ε, πρέπει να υπάρχει μια εσω... Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η εσωτερική αντίφαση όπως βλέπετε στην επιχειρηματολογία. Άρα το ερώτημα για τη δημοσιονομική ουδετερότητα είναι ανοιχτό και αξίζει να συζητηθεί περαιτέρω. Κατανοώ ότι το θέμα της διάρκειας θα συζητηθεί όσον ε, ούπο και όταν ε, έρθετε σε αυτό το θέμα θα πάρω πάλι το λόγο για να σχολιάσω. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, οι ίδιοι πόροι δεν έχουν ως στόχο να ξεφύγουμε από την τυραννία της δίκαιης επιστροφής και την ανάδειξη βεβαίως του κοινοτικού πνεύματος, της κοινοτικής μεθόδου, έτσι δεν είναι. Η ομάδα Μόντι αναφέρει ότι αν έχουμε ίδιος ιδίους πόρους, δηλαδή φορολογικές επιβαρύσεις που ε, τροφοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει σε αντιστάθμισμα οι φόροι σε εθνικό επίπεδο που επιβάλλονται να ελαφρυνθούν. Τέλος πάντων, πρέπει να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Ο κύριος Όλμπριχτ. Δεν είναι συμπέρασμα γιατί η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν έκανε μία συζήτηση. Απλώς ε, κλείνουμε εδώ αυτή την ε, συζήτηση και βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Και από αυτή τη συζήτηση προκύπτει ότι υπάρχει μια πρόταση από τον ε, ή τους εμπειρογνώμονες να μην αλλάξουμε την δομή του προϋπολογισμού κυρίως, αλλά να περάσουμε στο περιεχόμενο και να αλλάξουμε το περιεχόμενο. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί, αν δεν αλλάξουμε τη δομή, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς μας λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα πρέπει να περάσουμε στις, στους τομείς του προϋπολογισμού είτε θα σπάντων σε μεγάλα κεφάλαια, ας πούμε, στις επενδύσεις ή θα κρατήσουμε την ίδια λογική που έχουμε σήμερα και αν ναι, ε, το, τον καταλαβαίνουμε τον προπολογισμό. Το ερώτημα είναι βασικά, πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε βασικές ουσιαστικές αλλαγές. Στο Κοινοβούλιο συζητάμε τις νέες προτεραιότητες. τη σημασία που έχουν οι νέες προτεραιότητες. Κατά την άποψη των εμπειρογνωμών, οι νέες προτεραιότητες δεν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη φιλοσοφία. Απλώς πρέπει να αλλάξει την αποτελεσματικότητα και τις αναλογίες του προπολογισμού. Το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε τη δομή χωρίς να συζητήσουμε το περιεχόμενο. Merci. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ ένα σημείο. Ότι πρέπει να πλουστεύσουμε ουσιαστικά. Και δεν μιλάμε για τον ε, δημοσιονομικό προϋπολογισμό που συζητείτε, που θα βοηθήσει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιό να κάνει προτάσεις για το επόμενο πουδουπού, αλλά να υπάρξει και μια βαθιά μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού. Γιατί μας είπαν ότι δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε περαιτέρω τον τρέχοντα κανονισμό. Γιατί ε, είμαστε σε φάση εκτέλεσης του τρέχοντος που που. Εάν σε τρία χρόνια δεν μπορούμε να αλλάξουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο γιατί το υιοθετήσαμε πριν τρία χρόνια, ε, μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο. Επομένω, απλούστευση είναι το πιο βασικό από όλη απλούστευση. Έχουμε 40 λεπτά καθυστέρηση και πάμε στη δεύτερη στο δεύτερο γύρο συζητήσεων. Αλλά βλέπετε πόσο ενδιαφέρον προκάλεψε, προκάλεσε η πρώτη συζήτηση. Ο κύριος Άκος θα μας παρουσιάσει ένα, μια σύνοψη της μελέτης του για τη διάρκεια του επόμενου πουδουπού. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε πίεση χρόνου, λοιπόν θέλουμε να φύγουμε και οι δύο έχουμε αεροπλάνα. Θα προσπαθήσω να περιορίσω την παρέμβασή μου. Να μιλήσω το πολύ 15 λεπτά. Μετά από αυτή την ε, ενδελεχή συζήτηση για τη δομή και το περιεχόμενο του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ανάλυση για τη διάρκεια του ιδίου. Πριν όμως περάσω στην κάθε αυτό παρουσίασή μου, θέλω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλω να συνεισφέρω σε αυτή τη γενική συζήτηση για, το, για τη μελλοντική δομή του προπολογισμού. Μετά από την γενική συζήτηση θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε τρία σενάρια. Πέντε χρόνια, εφτά χρόνια ή δέκα χρόνια, δηλαδή πέντε συν πέντε το τελευταίο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Όλα θα τα συνοψίσουμε. Θα μιλήσουμε για την προβλεψιμότητα, τη σταθερότητα και από την άλλη την ευελιξία και την ανταπόκριση στις αλλαγές του προϋπολογισμού. Επιπλέον, θα ήθελα να μιλήσω για τα πρακτικά θέματα της εφαρμογής και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Μπορεί να μην έχω βέβαια αρκετό χρόνο για να μιλήσω και για το θέμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αλλά υπάρχει στην, ε, στο τέλος της παρουσίασής μου και στο τέλος της ε, μελέτης που έχετε σε υπόθεμα χαρτιού. Λοιπόν, καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια, μια γενική παρατήρηση καταρχήν. Θα ήθελα να καταλήξω ότι τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται. Έχουν συνηθίσει, μου λέει η εμπειρία μου, την εφταετή περίοδο του Πουδουπού. Και δεν τους ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Του ενδιαφέρουν τα τεχνικά θέματα. δύο, 2, συν 3 και κάποια άλλα τεχνικά θέματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την καθαρή δημοσιονομική θέση. Μάλιστα, δεν υπάρχουν λεπτομερείς μελέτες που έχουν ετοιμάσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ούτε το Κοινοβούλιο ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της διάρκειας. Υπάρχουν απλώς κάποιες παράγραφοι, κάποιες σύντομες αναφορές στο θέμα της διάρκειας του Πουδουπού. Στο πρώτο κομμάτι θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Για τα γενικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη παρατήρηση. Έχουμε ένα σύστημα λήψης των αποφάσεων που είναι τεχνοκρατικό και γραφειοκρατικό και βασίζεται σε κανόνες. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει δηλαδή ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κανονικά αυτή θα ήταν μια διαδικασία που γίνεται σταδιακά. Οι τομεί, οι γραμμέ του προπολογισμού μπορούν να μεταρρυθμιστούν, αλλά όχι μονομιά, βαθμιδών. Παραδείγματο χάρη, στο τρέχον ε, πουδουπού, Παρότι έχουμε σημαντικ... κάποιες σημαντικές αλλαγές, ακόμα και σήμερα το 72% των δαπανών δαπανώνται για την πολιτική συνοχή και τη γεωργική πολιτική. Η δεύτερη γενική παρατήρησή μου είναι ότι ο ενωσιακός προϋπολογισμός είναι ένας ε, προϋπολογισμός ε, επενδύσεων. Έχει διαφορετικές λειτουργίες από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μπορούμε να κοιτάξουμε Επιμέρου στοιχεία. Το βλέπετε στη μελέτη μου, βλέπετε την κλασική λειτουργία ενός προϋπολογισμού και κάνω τη σύγκριση και καταλήγω ότι ο ενωσιακός προϋπολογισμός ουσιαστικά κάνει μια ανακατανομή, γιατί η πολιτική συνοχής και μέρη η γεωργική πολιτική αφορούν την αναδιανομή πλούτου. Και υπάρχει και μια αναπτυξιακή λειτουργία. Γιατί και δύο αυτές πολιτικές, γεωργική και ε, συνοχής, αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές, ε, ε, διευρωπαϊκά δίκτυα, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη. Και αυτές οι πολιτικές συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης ανταγωνιστικότητας. Σε σχέση με την κλασική θεωρητική λειτουργία, την μακροοικονομική σταθεροποίηση, θα έλεγα ότι λόγω του μεγέθους του και μόνο του προπολογισμού αυτού, ο ενωσιακός προπολογισμό δεν είναι κατάλληλος για να εξασφαλίσει τη μακροοικονομική σταθεροποίηση. Προφανώς, κάποιες αλλαγές θα μπορούσαν να συμβούν στο μέλλον, πιο μακροπρόθεσμα, λόγω της μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής ε, μακροοικονομικής διακυβέρνησης. Θα ήθελα να μιλήσω για τα αμοιβαία ωφέλη των ε, μεταφορών πιστώσεων από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Βασικά πρόκειται για επανάληψη εν μέρη. Έχουν συζητηθεί αυτά τα πράγματα. Ε, η βασική καθαρή δημοσιονομική θέση είναι παραπλανητική. Είναι απλώς ένα στοιχείο των πλεονεκτημάτων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προφανώς υπάρχουν διάφορα αμοιβαία ωφέλη λόγω διασυνοριακών επιπτώσεων και μέσων επιπτώσεων στην ε, αγορά και την προσφορά και στη ζήτηση, συνέργεια, οικονομίες κλίμακας κτλ. κτλ. Εμείς, δηλαδή τα κράτη-μέλη ουσιαστικά, θα πρέπει να έχουν μια πιο ανοιχτή προσέγγιση και να μην εστιάζουν στενά στην καθαρή δημοσιονομική θέση. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Μήπως θα μπορούσατε να συνοψίσετε τη γενική προσέγγιση και να περάσουμε λιγάκι στη διάρκεια. Ναι, ναι, βεβαίως. Να πω δύο λόγια για τις επιδόσεις και την αιρεσιμότητα και τους σχετικούς κανόνες και την προστιθέμενη αξία, τα οποία τα αναφέρουν οι γενικέ μου παρατηρήσεις. Δεν θέλω να πω σε πολλέ λεπτομέρειες. Θέλω να καταλήξω ότι η προστιθέμενη αξία θα πρέπει να είναι στο κέντρο του ενωσιακού προπολογισμού και η αιρεσιμότητα θα πρέπει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, διότι υπάρχει μια σαφή σχέση ή θα πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στις μεταφορές πιστώσεων και στην συμμόρφωση βασικών μικροοικονομικών προϋποθέσεων και διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Και τέλος, μεγαλύτερη σταθερότητα και ευελιξία είναι και αυτά προφανώς εκ των ονουκάνευ. Αυτά είναι οι γενικές παρατηρήσεις τώρα. Μετά από αυτό το γενικό κομμάτι, θα ήθελα τώρα να περάσουμε στα τρία σενάρια. Έχω βάλει τους πίνακες αυτούς για τα τρία σενάρια. Ο πρώτος πίνακας μιλάει για τα θετικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα αρνητικά του πενταετούς πουδουπού, καταρχάς τα πλεονεκτήματα αυτού του σενάριου η ευθυγράμμιση με την εκλογική εντολή που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη θητεία της Κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κομισιόν και κάθε Κοινοβούλιο, ας πούμε, θα παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την προετοιμασία και την εκτέλεση και την εφαρμογή ενός πενταετούς πουδουπού. Αυτό σημαίνει ότι ο νοσιακός προπολογισμό και όλα τα συναφή θέματα και όλες οι συζητήσεις θα είναι στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών. Θα υπάρχει ως θέμα μονίμως και θα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα είναι μονίμως στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Το επόμενο πλεονέκτημα θα είναι ότι θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολότερη προσαρμογή σε απρόβλεπτα και σε αλλαγές. Η κασία είναι στην πραγματικότητα. Γιατί από την άλλη αυτή η ευελιξία θα εξασφαλιστεί μόνο με μεσοπρόθεσμα. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει προσαρμογή μετά και την πενταετία, την πρώτη, ας πούμε, τα πρώτα πέντε χρόνια. Ούτω ή άλλω θέλω να πω ότι απλούστεροι και πιο ευέλικτοι κανόνε είναι κάτι το απαραίτητο. Και θα προκύψουν και ω συμπέρασμα, ω αποτέλεσμα τη ε, βραχύτερη διάρκεια. Αν έχουμε απλούστερου κανόνε, θα είμαστε και πιο γρήγοροι στην εκτέλεση, για να μην έχουμε καθυστερήσει. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά χαρακτηριστικά του πεντέτου σπουδουπού. Φυσικά, βραχύτερη διάρκεια σημαίνει μικρότερη προβλεψιμότητα, ενδεχομένω. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πιο μακροπρόθεσμα. Για πιο μακροπρόθεσμε πολιτικέ, για πιο μακροπρόθεσμες επενδύσει. Παραδείγματο χάρη στην πολιτική συνοχή, στι υποδομέ πολιτικές για την έρευνα και ανάπτυξη, εκεί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα για τον πολιτή, ας πούμε, προγραμματισμό. Ένα άλλο αρνητικό χαρακτηριστικό θα είναι οι μόνιμες διαπραγματεύσεις που θα έχουμε. Από τη μία είναι και πλεονέκτημα, όπως σας είπα, από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι τα θεσμικά όργανα θα είναι σε μόνιμη διαπραγμάτευση. Κάτι άλλο αυτή η κασία για μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό εξαρτάται από τους κανόνες. Μέσα στην πενταετή διάρκεια δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα εξασφαλίσουμε αυτόματα μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη ευελιξία στον προπολογισμό. Τελευταία παρατήρηση για τα αρνητικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου πουδουπού, ενός πενταετούς δηλαδή πουδουπού. Θα έχουμε λίγο χρόνο για την προετοιμασία του επόμενου πουδουπού δηλαδή το δεύτερο χρόνο της εφαρμογής ε, ενός πενταετούς πουδουπού, θα πρέπει να ξεκινήσουμε στην πραγματικότητα την προετοιμασία του επόμενου. Χωρί καμία αξιολόγηση εξπόστα, εκ των υστέρων δηλαδή, χωρίς καθόλου αποτελέσματα για το τι πετύχαμε με το τρέχον πουδουπού, θα πρέπει να περάσουμε στην προετοιμασία του επόμενου. Το επόμενο πουδουπού λοιπόν θα βασίζεται στο που πουδουπού και όχι στο τρέχον. Το επόμενο σενάριο. αιτία. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει. Έγινε ο κανόνας. Είναι εποφελές για ένα πολιετή σχεδιασμό. Υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε σχέση με την πενταετία μπορεί να διευκολύνει πιο μακροπρόθεσμο και πιο στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι καλό για τις βασικές πολιτικές, για τους βασικούς τομείς παρέμβασης. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή και την αξιολόγηση. Τα αρνητικά όμως χαρακτηριστικά τώρα. Η εφταετή περίοδος δεν ευθυγραμμίζεται με την πενταετή εντολή που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα. Η Κομισιόν δηλαδή, η οποία ξεκινάει ένα εφταετές ας πούμε πουδουπού, έχει το σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία. Λόγω της ενδιάμεσης αναθεώρησης, η επόμενη Κομισιόν και το επόμενο Κοινοβούλιο βέβαια θα παίξουν και αυτά κάποιο σημαντικό ρόλο, αλλά διαφορετικό από τις προηγούμενες Επιτροπές και Κοινοβουλίου. Επίσης μπορούμε να το επικρίνουμε λόγω κάποιων ακαμψιών. Μπορεί να είναι αργός στις αντιδράσεις του. Δεν γίνονται γρήγορα προσαρμογές στα νέα δεδομένα. Γι' αυτό ακριβώς η ενδιάμεση αναθεώρηση είναι απολύτως απαραίτητη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση όπως ε, συνέβη και στην ε, περίπτωση του παρόντος ε, Πουδουπού βασίζεται μόνο στην εμπειρία που έχουμε από τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογή. Γιατί ξέρετε ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση πρέπει να προετοιμαστεί την τρίτη χρονιά. Και οι αλλαγές στους κανόνες θα πρέπει να περάσουν το πρώτο μισό του τέταρτου χρόνου της αυταετίας, έτσι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε μόνο μια διετή εμπειρία, ε, δεν είναι και πάρα πολύ Μπορεί να υπάρξουν και κάποιες καθυστερήσεις, κάποια προβλήματα. Λόγω των περίπλοκων κανόνων. Όπως ας πούμε για την πολιτική συνοχή. Συνέβη κάτι τέτοιο. Και δεν έχουμε πράγματι συσσωρευμένη εμπειρία για την ε, σωστή ενδιάμεση αναθεώρηση. Πάμε στο δεκαετές τώρα, ε, ε που, που. Καταρχάς, τα θετικά του. λόγω του χαρακτήρα της πενταετίας, 5 συν 5 δηλαδή, επίσης θα ευθυγραμμίζεται με τις εντολές που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα Κομισιόν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ υπάρχει ομοιότητα με, την, με το πρώτο σενάριο. Θα είναι όμως ε, μόνιμη προτεραιότητα για τα θεσμικά όργανα. Ε, θα δώσει όμως σταθερότητα, προβλεψιμότητα και κάτι πολύ σημαντικό, καλύτερη συμμόρφωσα με τις απαιτήσεις του στρατηγικού σχεδιασμού. Σημαίνει ότι θα έχουμε μία δεκαετία και κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τη δεκαετία. Κάτι που ξεκίνησε με τη στρατηγική της Λισαβόνας, μετά συνεχίστηκε με την Ευρώπη του 2020. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε την πρόβλεψη ότι μετά τη στρατηγική Ευρώπη 2020 θα περάσουμε σε μια στρατηγική για την Ευρώπη 2030. Για την επόμενη δεκαετία λοιπόν. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό και μια στρατηγική προσέγγιση. Αυτό τι σημαίνει. Ότι αν έχουμε ένα δεκαετές πουδουπού, όλες οι στρατηγικές, για μεγάλες στρατηγικές όπως το Ευρώπη 2020, ευθυγραμμίζονται με τη διάρκεια του πουδουπού. Μιλάω για διάφορες στρατηγικές, για την εκπαίδευση, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, για την έρευνα και την ανάπτυξη και για άλλε πολιτικέ. Βιώσιμη ανάπτυξη για θέματα που σχετίζονται με το κλίμα κτλ. Θα είχαμε πιο πολύ χρόνο για την συλλογή δεδομένων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή γιατί η ενδιάμεση αναθεώρηση βασίζεται ε. ουσιαστικά στα τρία πρώτα χρόνια της εφαρμογής, της υλοποίησης. Άρα θα είμαστε σε καλύτερη θέση σε σχέση με σήμερα σε ό,τι αφορά το επτάετες πω, σε ό,τι αφορά τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Η Επιτροπή με δεκαετές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αντιδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην όλη διαδικασία. Προφανώς. Το πραγματικό ερώτημα και αυτό αποτελεί την πραγματική απάντηση στο σενάριο για τα 5 συν 5 έτη είναι ότι τα νομικά μέσα και εργαλεία θα πρέπει να έχουν δεκαετή διάρκεια, το οποίο θα οδηγήσει σε κάποια α, έλλειψη ευελιξίας και αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, κάποιες αναθεωρήσεις που θα προβλέπονται. Θα πρέπει να βρούμε νομικά πώς θα λύθμισει το θέμα αυτό. Πρακτικά αυτό θα σήμαινε ότι σε κάθε κεφάλαιο θα υπάρχουν κάποια περιθώρια, κάποια αποθεματικά και επιπλέον σε ό,τι αφορά το σύνολο του προπολογισμού θα πρέπει να υπάρχει ένα σημαντικό αποθεματικό προκειμένου να δράσουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε ό,τι αφορά την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Μπορείτε να δείτε και το χρονοδιάγραμμα. Είναι ενδιαφέρον από πλευρά ε, πολιτικών κύκλων και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της ε, υλοποίησης ε, του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου στην περίπτωση των ε, σενάριων αυτών. Αυτό που είναι αρκετά ευαίσθητο είναι το χρονοδιάγραμμα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι συζητήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από κάποια συγκεκριμένη επιτροπή. Αλλά η εφαρμογή και τα συμπεράσματα θα είναι ουσιαστικά σε μια άλλη επιτροπή σε ένα άλλο κοινοβούλιο, σε μια άλλη θητεία. Θα σταματήσω το σημείο αυτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Και να ζητήσω από του εισηγητέ, έναν από του δύο εισηγητέ, την κυρία Τωμά να πάρει Σας ευχαριστώ πρόεδρε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκρίνηση αυτή. Πριν κάνω τις ερωτήσεις μου, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, γιατί αν σωστά κατάλαβα, αυτό που λέτε είναι το εξή. Η διάρκεια, το θέμα της διάρκειας, το είπε και ο κ. Ντεπρέ, δεν θα αποτελέσει το λόγο αντίστασης, αν θέλετε, από πλευρά του Συμβουλίου γιατί αυτό το θέμα ενδεχομένως να μην έχει μεγάλη πολιτική σημασία για το Συμβούλιο. Το αντίθετο πιστεύω και μάλιστα βρήκαμε και δυσκολίες ε, στο Συμβούλιο το, τη στιγμή που είπαμε ότι θα υπήρχε δυνατότητα αναθεώρησης στα πλαίσια της περίοδου 2014-2020 είδαμε πόσο απρόθυμο ήταν το Συμβούλιο και όταν θέλαμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση πάει ένας χρόνος τώρα και τότε πραγματικά καλέστε μας υποστηρίζει. Γιατί, γιατί πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά. Γιατί πρόκειται για μία δημοκρατική, αν θέλετε, διάσταση, μία ενωπητική διάσταση σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση αυτή, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση, σε ό,τι αφορά το πολιτή δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό οδηγεί και θα οδηγήσει τα κράτη-μέλη στην αντίσταση στις προτάσεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις προτάσεις αυτές. Θα είναι δύσκολος ο αγώνας. Είμαι ωστόσο απόλυτα πεπισμένη. Και αυτό φαίνεται και από τις τρεις προτάσεις και από τα τρία συστήματα που μας προτείνετε. Σας ευχαριστώ που κάθε φορά ε, παρουσιάζετε τα θετικά και τα αρνητικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε κάθε σενάριο. Εμένα, εγώ υποστηρίζω το 5 συν 5. Έτσι το 10 αν θέλετε έτη με υποχρεωτική αναθεώρηση στα 5 έτη. Είτε το κοιτάξουμε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, είτε το κοιτάξουμε σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει παράλληλα και να σεβόμαστε τους δημοκρατικούς κανόνες σε ό,τι αφορά την ανανέωση του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπής κάθε πέντε χρόνια. Αυτό φυσικά είναι απόλυτα απαραίτητο. Και θα πρέπει επίσης να βρούμε μια επαρκή χρονική περίοδο. Όχι μόνο για να υλοποιούνται οι πολιτικές και κυρίως τα θέματα τα διευθυντικά και να έχουμε υπόψη και το ιδιαίτερο περιβάλλον, γιατί υπάρχει το θέμα του περιβάλλοντος, του οικολογικού, της εργασίας, όπου απαιτείται προβολή και μακροπρόθεσμος χαρακτήρας και απ' την άλλη έχουμε άλλα ζητήματα στα οποία απαιτείται ευελιξία. Άρα θέλω μακροπρόθεσμη περίοδο, αλλά με υποχρεωτική, το τονίζω αυτό, είναι υποχρεωτική αυτή η αναθεώρηση. Όχι, πάει το review πέθανε. Division, Να μπει στο κείμενο. Κάτι υποχρεωτικό. Και φυσικά ανακύπτει άλλο ένα πρόβλημα στη συνέχεια. Αυτό το οποίο θα το αναθεωρήσουμε. Μάλλον τι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και τι θα πρέπει να παραμείνει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Γιατί άμα είναι να τα θεωρούμε όλα, ε, τι να μιλάμε για 10 χρόνια περίοδο τότε. Αν ε, από την άλλη η αναθεώρηση είναι περιθωριακή και πολύ ωριακή, γιατί να μιλάμε για 5 συν 5 έτη. Άρα, το θέμα είναι ότι αυτό που θα πρέπει να διαρκέσει ε, πολύ είναι διαρκή όσο χρειάζεται, αλλά να γίνεται εξωστή αναθεώρηση. Είχα θέσει και ένα ερώτημα στην προηγούμενη προγνώμονα, δεν μου απάντησε, γιατί επανέλθουμε στο, στο σκέλος της ευελιξίας. Τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις εξωτερικές κρίσεις, τα εξωτερικά αναπάντεχα συμπάντα. Εδώ δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για διάρκεια χρονική, αλλά και για μέσα ευελιξίας. Πέρα λοιπόν από την αναθεώρηση αυτή κάθε πέντε χρόνια, έχουμε και τα μέσα ευελιξία τα οποία μας επιτρέπουν να δράσουμε. Άρα, εγώ είμαι πεπισμένη απόλυτα για αυτό το 10-5 5 στην αναθεώρηση, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Το θέμα είναι τι θα πρέπει να περάσει από αναθεώρηση, τι θα πρέπει να μπορεί να θεωρηθεί και τι θα πρέπει να παραμένει απαράλλαχτο. Νομίζω ότι όμως η, ίδια, η πολιτική άσκηση της αναθεώρησης ε, είναι κάτι το απολύτω απαραίτητο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τωμά, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στο σκιό εισηγητή. Στον κύριο Λεβαντόφσκι. Uh, Κοιτάξτε, το θέμα της διάρκειας ε, έχει αναβαθμιστεί από την παραδοσιακή, αν θέλετε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου, ότι θα πρέπει το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο να συνάδει με τη θετία. Άρα πέντε χρόνια και όχι επτά. Το δικό μου θέμα είναι το εξή. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοια αντιστοιχεία γιατί το πραγματικό πολιτιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ε, προγραμματισμό, ό,τι και να λέμε, 5, 7, 5, 5 έτη, πάντα έχουμε κάποιους άγνωστους παράγοντες, όπως η διάρκεια των διαπραγματεύσεων. μισή χρόνια την προηγούμενη φορά. Πάνω από ένα έτος την προηγούμενη φορά. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε κάποιους μήνες ε, για το κατά πόσον θα διαρκέσει αυτή, πόσο, για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Και είχαμε και τα αναπάντηχα σήματα. Την προηγούμενη φορά είχαμε το Brexit. Τώρα έχουμε το Brexit. Πάντα λοιπόν έχουμε κάτι απρόβλεπτο. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική αντιστοίχηση. Πραγματική αντιστοιχία χρονική. Για να μην έχουμε λοιπόν ψευδεσίσεις να διαγράψουμε επιτέλους αυτή την παραδοσιακή αντίληψη του Κοινοβουλίου από τα χαρτιά μας. Στα επτά χρόνια ήταν πάντα λοιπόν η περίοδος αυτή και η ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να γίνεται όχι πάρα πολύ σύντομα, αλλά τουλάχιστον μετά από τρία χρόνια. Πέντε συν πέντε. αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα. Θα βρεθούμε σε αχαρτογράφικτα ύδατα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει εκ των προτέρων μετά από συζητήσει να τα ορίσουμε αυτά τι αποτελεί σταθερό και αμετάβλητο για 10 χρόνια και τι θα μπορούσε να μεταβληθεί και να μεταφερθεί. αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να εγκαταλείψουμε αυτό το παραδοσιακό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, τα, την πραγματική αντιστοίχηση τη θητεία με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Αν θέλουν οι σκιώδει να πάρουν το λόγο, κύριε κύριος Ντεπρέ. Ναι, εν συντομία κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να γίνει, να γίνει δογματικός στο θέμα αυτό. ακούγοντας και εσά και τους συναδέλφους ότι έχω να πω το εξή. Σε ό,τι φορά τα πέντε έτη αυστηρά, εγώ θα έλεγα όχι. Πέντε συν πέντε ενδεχομένω ναι. Σε ό,τι αφορά τα επτά χρόνια, θα έλεγα μάλιστα. Και θα εξηγήσω. Θα εξηγήσω γιατί. Γιατί αν ναι, είναι να πληρώσουμε κάποιο τίμημα για να αλλάξει αυτή η περίοδος, δεν βλέπω γιατί να το κάνουμε, ενώ πιστεύω ότι για να διατηρηθεί η ίδια διάρκεια, αν μπορούμε να επικεντρωθούμε σε τρία στοιχεία, θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά παραπάνω. Καταρχάς, μεγαλύτερη ευελιξία, σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία. Κατά δεύτερον, μείωση η μείωση του earmarking και κατά τρίτον να ορίσουμε το τι τους όρους υπό τους οποίους θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει αναθεώρηση. Αν μπορούσουμε λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το earmarking, σε ό,τι αφορά να... τις α, ε, συνθήκες αυτές και τους όρους αυτούς, εγώ ειλικρινά δεν θα ξεκινούσα μου για το πόσο θα διαρκέσει το πολιτεστημοσυνικό πλαίσιο, ειλικρινά όχι. Μάλιστα, ο Πρόεδρος θέλει Άλλο από τους κύριου εισηγητές να πάρει το λόγο. Μάλιστα, οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ. Δεν ναι, ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά μια και το συζητάμε, αισθάνομαι την ανάγκη να πάρω το λόγο. Νομίζω ότι είναι σαφέ ότι δεν πρόκειται να αποφασίσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Και προφανώ θα εξετάσουμε τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Ευελιξία, βεβαίω. Δεν χρειάζεται να το αναπτύξω αυτό. Όχι, ο κ. Φράντς δεν θέλει να πάρει το λόγο. Τον βλέπω και θέλει να πάρει το λόγο. Για τα πέντε χρόνια. Μα πες ότι συμφωνείς μαζί μου, λέει ο κ. Ο κ. Ένα πολύ σύντομο ερώτημα στον ειδικό μα τον εμπειρογνώμονα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση. Το πέντε, χρόνια παίρνει χ. Πρέπει να το απορρίψουμε και μας δώσατε τα επιχειρήματα. Αν ήσασταν σύμβουλος πολιτικών, τι θα του συμβουλεύατε. Καταλαβαίνω θα μου απαντήσετε εξαρτάται από το τι θέλουν οι πολιτικοί. Καλώς, ναι, εξαρτάται από το τι θέλουμε. Ε, τη δική σας νόμη ρωτάω και ζητάω. Ποια λύση είναι η καλύτερη. Σύμφωνα με αυτό που εσείς, εσείς θέλετε ή αυτό που νομίζετε ότι εμείς θέλουμε. Εφτά χρόνια με, τις δικές, με τους δικούς μας όρους, λέει ο κύριος Ντεπρέ. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Η κυρία Τωμά, εν συντομία πράγματι, πρόεδρε, ήθελα να, να απαντήσω και στον κύριο Ντεπρέ για τα 7 χρόνια. Ποιο είναι το πρόβλημα με τα 7 χρόνια. Ότι και εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αναθεώρηση. Το είδαμε αυτό. Άρα, η περίοδο τελικά είναι ακόμα πιο σύντομη. Ενώ με το 5 συ 5 τουλάχιστον έχουμε 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια κάνουμε αναθεώρηση. Και άρα υπάρχει αρκετό χρόνο να εφαρμοστούν πολιτικές και να φανούν ορατά τα αποτελέσματά τους. Με τον κύριο Όλμπριχτ είδαμε τις δυσκολίες της αναθεώρησης στα 3,5 χρόνια. Πολύ καλά τι κάνατε και πολύ καλά τα κάνατε, λέει ο κύριος Ντεπρέ. Εντάξει, τώρα άμα είναι αυτό το θέμα να μας κάνετε κολπλιμέντα δεν ε, υπάρχει σοβαρότητα. Ο Πρόεδρος. Βλέπω ότι ο κύριος Φερνάντες θέλει το λόγο. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Τα πέντε χρόνια όχι. Τα επτά είναι κάτι που δουλεύει. Μπορούμε να το βελτιώσουμε με περισσότερες ε, ευελιξίες. Αν πούμε 5 συν πέντε, με ρήτρα αναθεώρησης, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι μένουμε στα 5, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το συν. Και να έχουμε... Γιατί ε, αλλιώς λέμε 10. Δεν λέμε 5 συν 5, λέμε 10. Λέμε 10 με αναθεώρηση. Τότε θα πούμε 10. Αν πούμε 5 συν 5 με αναθεώρηση, τι είναι η αναθεώρηση. Μπορεί και να αναθεωρήσει κατά ένα δις, κατά 500 δις, 500 εκατομμύρια. Τα 7 λοιπόν είναι θέμα ασφαλεία. τα 10 γιατί όχι, αλλά τότε θα πρέπει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία από τα 7 στα 10. Ο Πρόεδρος, επιτρέψτε μου να πω ότι το ζήτημα είναι ουσιώδες και υπάρχει θέμα δημοκρατικής νομιμότητας, πραγματικό θέμα. Εσείς ήσασταν εδώ πριν την ανέωση της θητείας το 2014. Εγώ εξελέγην το Μάιο του 2014 και όταν έφτασα εδώ μου είπαν ακούστε είναι πολύ απλό, ο προϋπολογισμός έχει γίνει, ε, μας δίδεται ένα κομμάτι κάθε χρόνο και έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι εύθραυστο, κάτι επικίνδυνο. Πώς μπορεί κανείς να εμφανίζεται στους εκλογείς του και να λέει μην ανησυχείτε γιατί ο προπολογισμό έχει ήδη αποφασιστεί για τα επόμενα δέκα δεν θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ της αναδιανομής. Ο κύριος Φερνάντες, ναι, αλλά υπάρχει πρόβλημα, Πρόεδρε, γιατί μια διαπραγμάτευση για ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να γίνει παίρνει περισσότερα χρόνια. Μπορεί ενδεχομένω να πούμε ότι θέλουμε και κοινοβουλευτική θητεία να κρατάει 10 χρόνια. Είναι θέμα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό, πράγματι. Κοιτάξτε, οι εξελίξεις στον κόσμο επιταχύνονται. Όταν ψηφίσατε το τελευταίο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μειώσατε τότε τις πιστώσεις για τη μετανάστευση. Αυτό δείχνει την εξαιρετική σας πρόβλεψη του 2014, πόσο φανταστικές προβλέψεις κάνατε. Μετά όμως υπάρχουν άλλες δράσεις που χρειάζονται πολύ περισσότερη ευελιξία. 80% του προπολογισμού έχει ήδη τεθεί κατά μέρος 14% γίνεται αναδιανομή και 6% για τα θεσμικά όργανα, κοινοβούλιο, συμβούλιο, επιτροπή, δικαστήριο, λεκτικό συνέδριο και το καθεξής. Άρα να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ αυτού που αναδιανομείται και εκεί να έχουμε πιο απλούς κανόνες για αυτό το 14% γιατί επί ξέρετε οι άνθρωποι το μόνο που κάνουν είναι νύχτα μέρα να προσπαθούν να κόβουν και να ράβουν από τα σχέδιά τους για να τα ταιριάξουν και να τα χωρέσουν κακήν κακό στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι αρνητική προσθέμενη αξία. Ας κάνουμε μια ρήξη με αυτή τη μεθοδολογία μπορεί να δημιουργεί δουλειά για την Επιτροπή ή για την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά είναι αρνητική διαφήμιση και αρνητική προσθέμενη αξία και ο κόσμος δεν το αντέχει άλλο πια. Λοιπόν, κύριε Ισηγητά, έχετε το λόγο για τα συμπεράσματα και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό και απλό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, πρόθεση μου ήταν να μην σας δώσω μόνο μία καλύτερη επιλογή, να παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε σενάριου. Εν πάση περιπτώσει, κατέστη σαφές ότι η επιλογή παριθμών 1 δεν είναι βιώσιμη λόγω της πολύ βραχίας διάρκειας αυτής. Όμως, η επιλογή 2 και η επιλογή 3 εξαρτώνται από τους κανόνες και την ευελιξία. Και προφανώς, και επειδή όπως τα ανέφερα ήδη, ο προϋπολογισμός ο κοινοτικός έχει κυρίως να κάνει με επενδύσεις και μάλιστα μακροπρόθεσμες επενδύσεις απαιτεί μακροπρόθεσμη προοπτική και μακροπρόθεσμη σταθερότητα και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι στην πράξη η νομική βάση μπορεί να αποφασιστεί για 10 χρόνια στην περίπτωση των διευρωπαϊκών δικτύων, στην περίπτωση της πολιτικής για την έρευνα, για την ανάπτυξη, για τη συνοχή, πιο βασικά Μπορεί να γίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαρκή εμπειρία να λανσάρει ε, μακροπρόθεσμα προγράμματα, μακροπρόθεσμες δράσεις. Και αν δείτε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους εν γέννη, παρόλο που δεν υπήρξαν ριζοσπαστικές αλλαγές, έγιναν κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάποιες αναομαδοποιήσεις, αναδιατυπώσεις. Ο πρόεδρος διακόπτη. Επιτρέψτε μου κύριε Σιγητά, δεν έγιναν αλλαγές, αλλά αφού δεν είχαμε μέσα, πολλαπλασιάσαμε τους δορυφόρους του προϋπολογισμού. Άρα είναι καλό να εγγράψουμε την ανάγκη ενός ενιαίου ευανάγνωστου εύληπτου προϋπολογισμού στο κείμενο, να έχουμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό και αυτό να είναι μια ανάγκη που να εκφράσουμε ξεκάθαρα. Ο εισηγητής, ναι, απολύτως συμφωνώ. Είναι θέμα κανόνων. 10, 15, 20% π.χ. έστω του δεκαετούς πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να πούμε δηλαδή ότι θα βάλουμε το 10, 15, 20% ενός πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που ε, εκτείνεται σε 10 χρόνια να τεθεί ως αποθεματικό και μετά την αναθεώρηση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού γιατί μπορεί να υπάρξει μια, ένα σχέδιο εθνικό αναπτυξιακό σε έκταση δεκαετίας, ε, συμφωνία εταιρική σχέσης, θέσπιση πολιτικών για τη συνοχή, αντίστοιχη χρηματοδότηση και το καθεξής και να έχουμε συγκεκριμένα όρια, σημεία αναφοράς με δείκτες που θα ορίζουν τη νομική βάση με παρακολούθηση, με αξιολόγηση μετά το πρώτο ήμιση ή εξαρτάται πάλι από το ποιους κανόνες θα διαμορφώσουμε, π.χ. στα τρία χρόνια εφαρμογής ή στα τέσσερα ή στα πέντε και μετά να γίνουν προσαρμογές και ε, τροποποιήσεις και ε, ε νέες ομαδοποιήσεις και νέα προτεραιοποίηση, νέα ιεράρχηση ακόμα και εντός του προγράμματος συνοχής. Εξαρτάται από τους κανόνες που θα συμφωνηθούν. Να μπει 10% ή 15% των πόρων σε ε, αυτό το αποθεματικό. Και αυτό που είπατε στην αρχή έχει να κάνει με το νομικό πρόβλημα σε σχέση με τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών από τη μία και του Συμβουλίου δηλαδή κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης αναθεώρηση Θα συμφωνήσουν ότι είναι καθήκον Επιτροπής και Κοινοβουλίου να κάνουν την αναθεώρηση ή θα πούνε ότι πρέπει η δική τους φωνή να ακουστεί στις συζητήσεις. Είναι νομικό ζήτημα και αυτό. Πώς θα λυθεί. Προφανώς, εγώ θα ήμουν υπέρ η ενδιάμεση αναθεώρηση να αποτελεί καθήκον μόνο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν στο συνολικό πλαίσιο για τη δεκαετία και μετά να πάρουν το λόγο τα θεσμικά όργανα. Ο Πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε η συζήτηση. Θα πρέπει κάποια στιγμή να εξαχθούν τα συμπεράσματα και δεν θα είναι εύκολο αυτό, διότι επί της ουσίας ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης, τι θέλουμε να κάνουμε με την Ευρώπη. Όλο αυτό αποτελεί μέρος των συμπερασμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Βερμεέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς είναι ένα ειλικρινά ανοιχτό ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω καμία προκατάληψη κανένας στερεότυπο και καμία προηλημένη ιδέα και απόφαση. Θέλω να σας ευχηστήσω την προσοχή ε, σε δύο-τρία στοιχεία που ίσως δεν σας έχουν απασχολήσει σήμερα το απόγευμα. Για παράδειγμα, αυτό το επικείμενο και επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι χαρακτηριστικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ή μήπως δεν είναι δεδομένων των πολύ εξαιρετικών συνθήκων και περιστάσεων της απόσυρσης μιας χώρας που ε, συμφέρει πολύ στον προϋπολογισμό. Ίσως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για το αμέσως επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο απαιτούν αυστηρή πειθαρχία, εξαιρετικές ε, συμβιβαστικές λύσεις που να μην θέλετε εσείς να προδικάσετε και να κατοχυρώσετε και να δεσμευτείτε σε αυτές για δέκα χρόνια. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει ένα προσωρινό πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο μετά και μετά να υπάρξει το επίσημο πλέον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο των 27 πλέον χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως αξίζει δηλαδή μια τέτοια ε, σκέψη. Και αν πάτε σε ένα ρυθμό 5 συν 5, δεύτερη παρατήρηση, ποια είναι ε, χρονικά η κατάλληλη συγκυρία να το ξεκινήσει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν έχετε 5 συν 5 τώρα, θα ξεκινάει πάντοτε το έτος 21. Ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα ξεκινά πάντοτε 18 μήνες μετά από ένα πρόσφατα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 15 μήνες μετά από μια ε, πρόσφατα εκλεγμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιλεγμένη. Αυτό θέλετε? Το ορίζεται, δεν μπορεί να αλλάξει μετά η χρονική συγκυρία κάθε πότε θα πέφτει η έναρξη της διαπραγμάτευσης. Ίσως θέλετε να έχετε εξαετή περίοδο έτσι ώστε τελικά να, να μεταστραφεί χρονικά και να συμπέσει στη μέση της θητείας Κοινοβουλίου και Επιτροπής, το πότε θα ξεκινήσει το επόμενο, δηλαδή πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο κάθε φορά και ίσως αξίζει αυτό να το εξετάσετε εξαετή περίοδο για αυτό το λόγο, για να σας συμφέρει χρονικά. Έχω σύν της άλλης εμπειρία 20 ετών στα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια και αυτό που έχω μάθει είναι ότι είναι ένα πακέτο. Κάθε στοιχείο, κάθε πολιτική, κάθε πρόγραμμα ε, έχει ένα κράτος μέλος που το στηρίζει και που το θέλει ή κάποιο μέλος του Κοινοβουλίου που το στηρίζει και που το θέλει. Άρα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε δύο κατηγορίες προγραμμάτων. Μία κατηγορία που θα έχει 10 χρόνια γραμμένα στο μάρμαρο που δεν θα μπορούν να αποτέλεσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μία δεύτερη κατηγορία προγραμμάτων που θα πάρει μόνο την πενταετία. Η ανησυχία μου είναι ότι από τη στιγμή που τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι ότου όλα συμφωνηθούν, ε, χρειαζόμαστε 10 χρόνια ε, πλήρως ε, συμφωνημένα τα 99,5% των πραγμάτων και η ενδιάμεση αναθεώρηση δεν θα μπορεί να αλλάξει τίποτα που έχει ήδη τεθεί κατά μέρο ω αποθεματικό ή έχει ήδη κατευθυνθεί σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα μπορούν να αλλάξουν μόνο κάτι φιωριτούρε πολύ επιφανειακέ. Αυτό δηλαδή με ανησυχεί. Από τη στιγμή που έχουμε το ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα, θα δυσκολευτούμε να κάνουμε ουσιαστικέ αλλαγέ με την ενδιάμεση αναθεώρηση. Όλες αυτές είναι οι σκέψεις που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, σας ευχαριστώ που προσθέσατε το τέταρτο σενάριο των έξι ετών. Περιμένω κάποιος άλλος να πλειοδοτήσει και να πει εννιά. Αλλά τουλάχιστον παραιτηθήκατε από τα τέσσερα χρόνια. Καλό είναι αυτό. Να δεσμευτούμε για δέκα χρόνια σε ένα κόσμο που αλλάζει τόσο πολύ, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχουμε συνάμα εργαλεία ευελιξίας, ακριβώς για να αποφύγουμε την ακαμψία η οποία θα αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας προτείνει trust fund, ε, καταπιστέματα, ταμεία και ένα γαλαξία εργαλείων και μέσων που δεν σημαίνουν τίποτα για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα της δημοκρατίας μας. Συμπερασματικά, Ποιο από του δύο εμπειρογνώμονε θέλει να πάρει το λόγο, από του δύο εισηγητέ, Η κυρία Τωμά τον θέλει περισσότερο από όλου τον λόγο. Παρακαλώ. Ναι, γιατί με τον κύριο Όλμπριχτ τα προβλέπουμε όλα πάντοτε εκ των προτέρων και είχαμε συνοηθεί ότι εγώ θα πάρω το λόγο τελευταία. Ακριβώ, στο σχόλιο εκτό μικροφώνου, απαντάει η κυρία Τωμά. Λοιπόν, καταρχά πρέπει, όπως έλεγα και προηγουμένως, να έχει κανεί υπόψη του το εξή. Αν δεχθούμε τα 7 χρόνια, τότε η ενδιάμεση αναθεώρηση θα γίνεται κάθε 3,5 χρόνια, άρα κάθε πιο σύντομη χρονική περίοδο από ό,τι τώρα ισχύει. Προσπαθούσα πριν να κάνω μια σύνοψη με τον κύριο Τεπρέλα, δυσκολεύτηκα. Το να πούμε ότι 5 συν 5 με ρήτρα αναθεώρηση και 10 από την άλλη με ενδιάμεση αναθεώρηση είναι σαν να λέμε το ίδιο πράγμα από δύο διαφορετικέ οπτικές γωνίες. Όλα εξαρτώνται από αυτά που θα βάλουμε στο κορβανά της υποχρεωτικής αναθεώρησης. Η πραγματική συζήτηση δεν είναι η διατύπωση, αν θα διαλέξουμε τις λέξεις 5 συν 5 ή 10. Η αληθινή συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ποιε είναι οι μακροπρόθεσμες πολιτικές που δεν θα αγγιχτούν, δεν θα αλλάξουν και ποιε είναι οι πολιτικές ακριβώς για να αποφύγουμε αυτό το... Ε, αυτό που έλεγε ο Πρόεδρος, τη δημιουργία των trust fund, των καταπιστευματικών ταμείων, για να έχουμε πολιτικές πραγματικά προστιθέμενης αξίας. Πρέπει να έχουμε ευελιξία, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε τη στιγμή της αναθεώρησης. Αυτή είναι η αληθινή συζήτηση. Άρα πρέπει να συζητήσουμε και για τις μακροπρόθεσμες πολιτικές που δεν μπορεί κανείς να τις αγγίξει και να τις αλλάξει, αλλά και τις πολιτικές όχι τόσο βραχυπρόθεσμες, αλλά που χρήζουν εν πάση περιπτώσει μεγαλύτερης ευελιξίας. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μας εφίστησε την προσοχή σε αυτό το ενδεχόμενο του μεταβατικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ήδη αλλιώ το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό να το βάλουμε στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, το προσωρινό μεταβατικό πλαίσιο, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και σας ευχαριστώ για τις προϋποθέσεις αναθεώρησης, το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να είναι πολύ καλά προσδιορισμένες και καθορισμένες όποια επιλογή τελικά και αν κρατήσουμε. Και θέλω να πω ότι ακόμα και στις μακροπρόθεσμες πολιτικές πρέπει εκεί να συμπεριλάβουμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα με την πολιτική συνοχή, για έστω. Αν αντιληφθούμε ότι δεν δουλεύει, θα την καταργήσουμε όχι, δεν την καταργούμε. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο την εφαρμόζουμε. Αυτό που δεν λειτουργεί, αλλά δεν πρέπει να καταργηθεί και αυτό πρέπει να μπορεί να γίνεται και να γίνει. Και τέλος, για να απαντήσω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν λέτε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε βραχυπρόθεσμες πολιτικές από τη μία και μακροπρόθεσμες από την άλλη, γιατί η διαπραγμάτευση είναι package, είναι πακέτο, τότε ας έχουμε ακριβώς μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πολιτικές, ακριβώς για να μην υπάρχουν πακέτα. Τι θα πει συνολική συμφωνία και τίποτα δεν έχει κλείσει μέχρι ότου να κλείσουν όλα. Θα πει να έχουμε τα rebate, τις επιστροφές, ε, τα, τις λύσεις ad hoc που είναι ε, ε, κοντόφθαλμες και τις οποίες θέλουμε να κάνουμε μια φυγή προς τα εμπρός, ένα άλμα να τις ξεπεράσουμε για να αποφύγουμε τέτοιου είδους τέτοιου είδους ε, ευρεσιτεχνίες. Πρέπει να σπάσει πλέον αυτό το απόστημα, θέλετε, αυτός ο μηχανισμός, αυτός ο κύκλος των ε, δικαίων επιστροφών και ούτω καθεξής. Εγώ έτσι βλέπω τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Όλμπριχ, θεωρείτε ότι έχετε καλυφθεί, όλα έχουν υποθεί. Θέλετε λοιπόν να ε, διασπάσετε, να καταγγείλετε και να καταστρέψετε πλέον την τυρενία της δίκαιης επιστροφής και γι' αυτό πρέπει να ασκήσετε ανήλαιη πίεση στον κύριο Λεβαντόφσκι και στους λοιπούς όσο περισσότερο εισφέρουν τα κράτη-μέλη, τόσο περισσότερο θα σταματήσουμε να μιλούμε για τη δίκαιη επιστροφή και θα αναδυθεί πλέον ένα πραγματικά κοινοτικό αλληλέγγυο ε, πνεύμα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει εξ αρχής. Καλώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα προχωρήσουμε γιατί οι διερμηνείς θα παραμένουν μέχρι τις 6.30 στην αίθουσα. Η κυρία Γκάρντια Θαμπάλ είναι έτοιμη να μας παρουσιάσει μια έκθεση που είναι κάτι το κενοφανές. Μια έκθεση δικιά μας της Επιτροπής στον Προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, είχα ετοιμάσει μια παρουσίαση εκτεταμένη και λεπτομερή της έκθεσης. Όμως, έχουμε καθυστερήσει μισή ώρας και γι' αυτό θα παρουσιάσω συνοπτικά μόνο τις βασικές γραμμές της έκθεσης αυτής. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά με τη νέα διαμόρφωση της Επιτροπής μας που έχουμε το καθήκον να συντάξουμε έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για να το πράξω προσπάθησα να συμπυκνώσω όλες τις ιδέες σε πέντε μεγάλα κεφάλαια, αν θέλετε, ή εδάφια. Πρώτον, κάνουμε μια ανάλυση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς σχετίζονται όλες αυτές με τις πολιτικές που υπερασπιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς σχετίζονται με τα project, τα προγράμματα, τα έργα, τις γραμμές επενδύσεων που ε, κάνει και η τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι βασικός παράγοντας που κινητοποιεί κρατικά κονδύλια αλλά και κονδύλια του ιδιωτικού τομέα για να γίνονται επενδύσεις. Και γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι πολιτικέ τη τράπεζα στηρίζονται στην ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών, στη στήριξη τη πραγματική οικονομία, στην αηφόρα ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, στήριξη τη καινοτομία, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στήριξη τη πολιτική συνοχή και είναι δίκαιο να τονίσει κανείς την καλή δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είναι δίκαιο να απαιτήσει να κάνει ακόμα περισσότερο και να στηρίξει περισσότερο τις χώρες που το χρειάζονται. Και να πάει στο όριο, να κατέβει στο όριο του τριπλού α από τη στιγμή που δεν της επιτρέπεται να κατέβει πιο κάτω, τουλάχιστον να το εξαντλήσει, να είναι μόνο ε, μία στιγμή ένα, μία μικρή γραμμίτσα πάνω από το τριπλό α στην αξιολόγησή της, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχει κινητοποιήσει όσο δυνατόν περισσότερο ε, κονδύλια για να στηρίξει αυτές τις χώρες. άλλο εδάφιο λοιπόν είναι η συμμόρφωση ε, και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αναθεωρήσει τη στρατηγική της για την ενεργειακή πολιτική και θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια για να εγκαταλείψει σιγά σιγά τη χρηματοδότηση της ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα και να χρηματοδοτήσει περισσότερο project, προγράμματα, σχέδια που βασίζονται σε καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Βεβαίως έχει ρόλο να διαδραματίσει στη διαχείριση της κρίσης και την ε, αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Υπάρχει πρωτοβουλία για την κατοικία, για τη μόνιμη παραμονή, για ε, την αηφόρο ανάπτυξη, για τα... είναι βασικός εταίρος για όλες αυτές τις πολιτικές. Άρα χρειάζεται καλύτερος και περισσότερος συντονισμός. Αυτό θα είναι κάτι θετικό. Ε, είναι παρούσα η τράπεζα και στην πολιτική για την ισότητα των φύλων. Έχει οθετήσει στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τώρα πρέπει να συντάξει σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων και έχει και ένα κοινωνικό πυλώνα, η Τραπεζή Επενδύσεων έχει ένα πυλώνα χρηματοδότησης υποδομών που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με την κατοικία, με ε, τα συστήματα υγείας μεταξύ άλλων. Αυτά λοιπόν. Ένα δεύτερο τμήμα στην έκθεσή μου έχει να κάνει με την Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα θέματα φορολογίας, φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και ούτω καθεξής. Φιλόδοξη πρέπει να είναι η πολιτική της σε σχέση με του, τα θεσμικά ιδρύματα που δεν συνεργάζονται. Πρέπει να κινητοποιεί περισσότερο το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, και είναι σε θέση να είναι πρωτοπόρος, να αναλάβει ηγετικό ρόλο, να αποτελέσει υπόδειγμα στην τροποποίηση των σχέσεων ή των μη σχέσεων με δικαιικά συστήματα και ένομες τάξεις που δεν συνεργάζονται ε, σε θέματα φοροδια... καταπολέμησης φοροδιαφυγής και φόρο αποφυγή. Πρέπει να απαιτήσουμε από την Τράπεζα Επενδύσεων να συντάξει εκθέσεις αναχώρα για να έχουμε καλύτερο και περισσότερο έλεγχο. Τρίτο τμήμα στην εκθεσή μου είναι η διαφάνεια, δεδομένου του μεγέθους των κονδυλίων που χειρίζεται, με το γεγονός ότι είναι όλο και πιο παρούσα στις ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Ο προπολογισμό, ούτω ή άλλω εγγυάται την εφαρμογή όλων αυτών των πολιτικών και εμεί θέλουμε διαφάνεια και διαβίβαση των εγγράφων επικοινωνίας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αποτελούν ε, ε, αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να είναι τόσο χαρακτηριστικά, η διαφάνεια για παράδειγμα, όσο το λογότυπό της και η ονομασία της και το όνομα με τον οποίο είναι γνωστή στην αγορά. Δηλαδή πρέπει να καταλήξουμε στο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ίσον διαφάνεια. Υπ' αυτή την έννοια, καλό θα είναι να συμπεριλάβουμε μια ιδέα που ακούσαμε για τα, ε, την περασμένη εβδομάδα με τα investment windows, τις επενδυτικές απευθυντικές ε, θηρίδες, ποιους στόχους ανάπτυξης ε, επιδιώκει ο καθένας, ποιους στόχους θέλει να πετύχει και γι' αυτό ζητά χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι θα εντάξουμε τους στόχους τους περιβαλλοντικούς και άλλους στα προγράμματα. Και πρέπει να ενεθωρηθεί και το σύστημα των, ε, της χρηματοδότησης. Τι σημαίνει, τι συμβαίνει, υπάρχει πρόβλημα μετάφρασης. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Συνεχίζει ο Μιλήτρια. Έχουμε λοιπόν το σύστημα των παραπώνων, των προσφυγών ε, και πρέπει να μεταρρυθμιστεί αυτό το σύστημα των προσφυγών έχει ασκηθεί κριτική και, στο από το διαμεσολαβητή και από άλλους. Πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική στον τρόπο με τον οποίο θα τροποποιήσουν το σύστημα προσφυγών ακριβώς για να ε, βελτιωθεί σημαντικά. Στο, στο τέταρτο τμήμα μιλώ για τις οικονομικές δραστηριότητες, τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αποσκοπεί στο κοινό όφελο, στο κοινό συμφέρον, στο κοινό δημόσιο καλό και να βελτιωθούν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις ορισμένων έργων και προγραμμάτων για να έχουν προστιθέμενη αξία και να συμβάλλουν με τις πολιτικές που υπερασπιζόμαστε ή να συνάδουν με τις συνθήκες της αγοράς σε κάθε χώρα. Γιατί το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε κάθε χώρα δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες, άρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να έχει μια πολιτική διαφοροποίηση των προϊόντων των χρηματοδοτικών που προτείνει για να προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις ιδιορυθμίες των εθνικών χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Και τέλος, μιλώ για τη συμβουλευτική και το συμβουλευτικό της ρόλο. Ξέρετε, πολύ συχνά οι τελικοί αποδέκτες δεν γνωρίζουν τα προγράμματα που τους διατίθενται και στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν. Πρέπει λοιπόν να αναλυφθεί ένας πιο ενεργητικός ρόλος στο τομέα των επενδύσεων, το της επικοινωνίας με συγχωρείτε, και πρέπει όλοι να αναλάβουμε αυτό το καθήκον, έτσι ώστε η επικοινωνία να είναι καλύτερη, να στηριχθούν ε, οι χώροι φορείς έτσι ώστε η πληροφορία να φτάσει σε όλους και να μην μείνουν κονδύλια αναξιοποιητά και να μην υπάρχουν έργα που δεν θα τύχουν χρηματοδότησης ή δανειοδότησης γιατί υπάρχει απουσία συμβουλευτική ή απουσία γνώσεων και πληροφορίες για την ύπαρξη του συγκεκριμένου δανείου χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Πολύ πλούσια η παρέμβασή της. Πολλά στοιχεία μας έδωσε. Δεν θα δεν ζητάω καν την αντίδραση του κυρίου Ολιβιέ από την τράπεζα. Θα σας το δώσω πρώτα αυτόν τον λόγο. Θα ζητήσω από τους κοιόδης ε, εισηγητές να πάρουν τον λόγο. Ο κ. Μορεσάντ, τηλεγραφικά. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια από τα θέματα τα οποία θα θίξω και τις τροπολογίες μου. Καταρχάς, ευχαριστώ την AIDER για την έκθεση που αναφίβολα κινείται προς αυτή κατεύθυνση και όταν λέω αυτό δεν είναι ότι εννοώ πως έχει κάνει μια δουλειά προς την κατεύθυνση και εμείς πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερη προσπάθεια για να τη συμπληρώσουμε. Όχι. Απλώς υπάρχουν κάποια επιμέρους σημεία που θα πρέπει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Καταρχάς το ΕΦΣΙ. Ε, η Τράπεζα Επενδύσεων συνεισφέρει πολύ στο Μα Θα πρέπει νομίζω να σταθούμε περισσότερο, με περισσότερες λεπτομέρειες στο ΕΦΣΙ στην έκθεσή μας. Διαλέξαμε στην περίπτωση του ΕΦΣΙ να χρηματοδοτήσουμε τα καλύτερα project, τα καλύτερα έργα, χωρίς γεωγραφική εκπροσώπηση. Δεν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, αλλά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση υπερβολική σε κάποια κράτη-μέλη. Γιατί τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, ειδικά σε κάποια νέα κράτη-μέλη, έχουν διαφθορτικά ελλείμματα. Δεν έχουν ε, πείρα από χρηματοδοτικά εργαλεία, πείρα γενικά. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να τους ε, παράσχει συμβουλές και τεχνική αρρωχή, ειδικά σε αυτά τα κράτη που έχουν ε, διαφορετικά ελλείμματα. Ε, υψηλό πιστοτικό επίπεδο. Είναι σημαντικό θέμα. Φυσικά θα θέλαμε η τράπεζα ε, να επενδύει σε καλά project αλλά και σε πιο επικίνδυνα ε, project. Δεν υπάρχει αντίφαση σε αυτό. Ξέρουμε, ξέρουν καλύτερα από εμάς, από, ε, ξέρουν καλύτερα συγγνώμη από εμάς για το πώς θα επενδύσουν το χαρτοφυλάκιο τους. τέταρτον, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεγαλύτερη εστίαση εκεί. Γιατί αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων απασχόληση και ξέρουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη οι μικρομεσαίε επιχειρήσει εξακολουθούν να έχουν δυσκολίε με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Για την, τον εξωτερικό δανεισμό και την εντολή σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να δούμε πώ θα το συζητήσουμε περισσότερο τι επόμενε εβδομάδε και θα το σχολιάσουμε στην έκθεση αυξανόμενος ρόλος για την ε, Τράπεζα Επενδύσεων, για την ε, μεταναστευτική κρίση και τους, ε, τις οδούς μετανάστευσης. Πήγαμε στην Τινησία, στο, στην Ιορδανία και το Λίβανο και η Τράπεζα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές, σε ενέργεια, σε ανεφοδιασμό σε είδωρ, αλλά υγεία, εκπαίδευση κοινωνικές υποδομές, ε, ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υποστήριξη τοπικών μικρών επιχειρήσεων. Τελευταίο σχόλιο, το Brexit. Το Brexit θα επηρεάσει τις δραστηριότητες της Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι προς το συμφέρον μας να υπάρξει μια συνέχεια στις δραστηριότητες της Τράπεζας. Μια ομαλή μετάβαση από την ε, Τράπεζα Επενδύσεων των 28 κρατών σε τράπεζα των 27 κρατών. Είναι σημαντικό αυτό. Και Έιντερ, θα συνεργαστώ και μαζί σου και με τους σκιώδεις συζητητές σε επόμενες εβδομάδες για το θέμα αυτό. Κύριο Σάλλη. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Συγχαίρω την εισηγήτρια καταρχήν για την ευρεία εμβέλεια της ε, έκθεσης. Ε, καλύπτει όλες τις αστριότητες της τράπεζας. Ε, παρουσιάζει τις ε, δράσεις, ε, όλες τις δράσεις της τράπεζας, χρησιμοποιητικές επιχειρήσεις, επικοινωνία, τα πάντα παρουσιάζονται. Είναι σωστή η προσέγγιση, γιατί ο ρόλος της τράπεζας είναι να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναπτυξιακά εργαλεία. Καταλητικός ρόλος της τράπεζας μέσω της χρηματοδότησης είναι βασικό στοιχείο για να καθοριστεί και να αυξηθεί η προστέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλιστεί ηγετικό ρόλο για την Ευρώπη στην ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, υποδομέ και ελκυστικότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τη σημασία τη συνέπεια στι χρηματοδοτικέ δραστηριότητε τη Τράπεζα με την ε, συνολική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πολιτικέ προτεραιότητε. Είναι βασικό παράγοντα για την αναθέρμανση τη ευρωπαϊκή οικονομία και τη αύξηση τη αποτελεσματικότητα των οικονομικών πόρων ε, συστηματικά θα πρέπει η τράπεζα να προσέχει μεσοπρόθεσμα και βαρχοπρόθεσμα τις επιπτώσεις όταν καθορίζει τις επενδυτικές της δράσεις και παίρνει αποφάσεις για αυτές. Ε, η ανάπτυξη του ΑΕΠ και η δημιουργία ε, ευκαιριών απασχόλησης είναι σημαντικό γι' αυτό. Θα πρέπει να ε, αξιολογήσουμε τις δράσεις της τράπεζας μέσω μιας μελέτης αντικτύπου. Ε, βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα μέχρι το 2017. Ε, επιπλέον 0,8 ε, σε ΑΕΠ και αύξηση των θέσεων απασχόλησης 30.000. Μέχρι το 2030 ε, θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4 και επιπλέον θέσεις απασχόλησης 1,4 εκατομμύρια. Θα ε, ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάκαψη στην Ευρώπη και κυρίως κάποιοι τομείς, κάποιες γεωγραφικές περιοχές θα πιάσουν τις πιο προστινές τι πιο πρωτοπόρε Είναι σημαντικό όμως να γίνονται επενδύσει σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, η επίπτωση της τράπεζας στην εφαρμογή των ε, βασικών δημοσίων πολιτικών μπορεί να παρακολουθείται μέσω των αποτελεσμάτων των επενδύσεων σε βασικούς τομείς. Η καινοτομία, ε, δεξιότητες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποδομές, περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα πρέπει να καθορίζει την, τους τη με βάση τη συνεισφορά στις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές των δρασιών της. Η ενθάρρυνση ε, προς την διαφάνεια της τράπεζας και τον εσωτερικό έλεγχο είναι προϋπόθεση για καλύτερη ε, εταιρική διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό η τράπεζα να συνεχίσει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής, παράτυπων ενεργειών και εξεπλήματος του χρήματος. Μην ξεχνάμε τη σημασία το χρημα... της χρηματοδότησης της τράπεζας. Είναι σημαντικό οι δραστηριότητε της να λαμβάνουν χώρα τηρώντας τα πιο αυστηρά πρότυπα. Ευχαριστώ. Δεν ζητάει κανένας άλλο βουλευτή το λόγο. Γι' αυτό ο κ. Ολιβιέ. Από την τράπεζα θα παρέμβει, αλλά σύντομα αν γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την παρουσίαση. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να αντιδράσω ε, για κάποια επιμέρους σημεία, σε κάποια επιμέρους σημεία σύντομα. Καταρχά ε, συμφωνούμε με τη γενική διάγνωση που γίνεται στην έκθεση και για την οικονομική ανάκαμψη και για την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Η ενθάρρυνση των επενδύσεων γίνεται ήδη, υλοποιείται ήδη. Αλλά υπάρχουν ανισορροπίε μεταξύ τομέων, χωρών και περιφερειών. Ξέρουμε την κατάσταση στι δημόσιε επενδύσει. Υπάρχει μια συρρήκνωση έντονη τη στιγμή της δημοσιονομικής ε, παγίωσης, ε, σταθερότητα, Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να ενθαρρυνθούν οι δημόσιε και ιδιωτικέ επενδύσει. Εκεί ακριβώ η τράπεζα μπορεί να συνεισφέρει και κάνει την προστιθέμενη αξία, κάνει τη διαφορά. Το επενδυτικό σχέδιο και η εφαρμογή του ΕΦΣΙ ήταν ένα βασικό στοιχείο, μια ατμομηχανή για την ε, δραστηριότητα της τράπεζας. Η τράπεζα μπόρεσε να ε, δραστηριοποιηθεί σε επιχειρήσεις υψηλότερου κινδύνου. Ε, ακριβώς αυτή είναι και η θέληση της τράπεζας να εξασφαλίσει ότι η, χρηματοδότηση εξασφαλίζει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Χρηματοδότηση τη τράπεζα δηλαδή. Λοιπόν, για τι προτεραιότητε τη τράπεζα, να αντιδράσω λιγάκι. Έχει σαν αποστολή να υποστηρίξει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, έτσι. Αυτό είναι προφανέ. Σε σχέση με την ανησυχία που υπάρχει για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι αν όχι ο νούμερο ένα στόχο, ένα από του βασικού στόχου τη τράπεζα. Αν κοιτάξτε τον όγκο των δραστηριοτήτων μα για το 2016, υπογράψαμε 86, ε, συμβάσεις 86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ε, και τα 33,4 δισεκατομμύρια ήταν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάσεις για τις μικρομεσαίες. Ε, είναι σημαντικές οι ελλείψεις αγοράς στον τομέα αυτό, γι' αυτό λοιπόν ένας θεσμός όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο. Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική ισορροπία υπάρχει μια θέληση πάλι από πλευράς τράπεζας και το επενδυτικό σχέδιο ήταν ένα κίνητρο για να δουλέψουμε περισσότερο με τις δημόσιες τράπεζες ε, και τις εμπορικές τράπεζες, ούτως ώστε να έχουμε σημαντική περιφερειακή επίπτωση και να αναπτύξουμε, την τεχνική αρρωγή. Γιατί είναι σαφές ότι όλα τα κρατημέλη δεν έχουν μια τέτοια τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει δομές και έργα. Η τεχνική αρρωγή με μια ενισχυμένη παρουσία σε τοπικό επίπεδο είναι για μας σημαντική στο βαθμό του δυνατού βέβαια η τράπεζα προσπαθεί να είναι παρούσα και φυσικός πώς, να υπάρχει, δηλαδή να έχει, ε, να έχει υποκαταστήματα είτε να έχει συνεργάτες ε, επιτόπου για να υλοποιήσει την τεχνική αρρωγή. Για το θέμα της ε, διαφάνειας τώρα που αναφέρθηκε και της ε, φορολογίας είναι προφανώς προτεραιότητα για την τράπεζα. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες μας ανάλογα με τα νέα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα φορολογικά και για τα θέματα διαφάνειας. Φερρυπίν, από τις αρχές του 2017 έχουμε αρχίσει να, ε, να δημοσιεύουμε τα πρακτικά των συζητήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μια πρώτη φάση. Φυσικά πάντα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Sur la communication. Για την ανακοίνωση, έχετε να πείτε κάτι επικοινωνία, συγγνώμη. Si je peux revenir Για την επικοινωνία. Προσπαθούμε να επικοινωνούμε περισσότερο για τα έργα που υποφελούνται από τη χρηματοδότηση της τράπεζας και, από την, και που στηρίζονται και από τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Είναι ένα θέμα που γνωρίζουμε, το έχουμε υπόψη μας. Η τράπεζα θα το δουλέψει περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Από τη Γενική Διάθεση Προπολογισμού κάποιες ε, παρατηρήσεις. Alors, Ποιο Τι θα πάρει το λόγο από την ΕΚΦΙΝ. Τα πιο πολλά σχόλια και οι πιο πολλέ συστάσει οι οποίε ε, περιλαμβάνονται στην ε, έκθεση στρέφονται και απευθύνονται στην ΕΤΕΠ. Οπότε δεν έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Σημειώνουμε τα σχόλια και την υποθέτηση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ΕΤΕΠ και θα παρακολουθήσουμε και τις τροπολογίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καρτίζα Βάλ θέλει να πάρει το λόγο για να συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ σύντομα γιατί βλέπω μέσω των πανεβάσεων των άλλων εισηγητών αλλά και του εκπροσώπου της τράπεζας ότι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Οι επιθυμίες μας για το μέλλον ε, ταυτίζονται. Μία εξήγηση θέλω να δώσω μόνο για δύο σημεία που ανέφερε ο κ. Μουρεσάν. Το ΕΦΣΥ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταρχάς, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για το ΕΦΣΥ. Θεωρούσαμε ότι είχαμε συμφωνία ήδη, αλλά είναι όλα λιγάκι στον αέρα. Νόμιζα ότι είχα χρόνο για τις τροπολογίες και για να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά ξέρετε ότι αυτές οι εκθέσεις πρωτοβουλίας ε, πιέζονται, ας πούμε, χρονικά. Τα αφήνουμε λιγάκι στον αέρα αυτά τα πράγματα, για το ΕΦΣΙ δηλαδή, και στη φάση των τροπολογιών θα τα συγκεκριμενοποιήσουμε. Επίσης, ε, για την πολιτική, ε, την περιφερειακή. Ε, την άποψη της Επιτροπής ε, Ρέτζι θα την ε, ενσωματώσουμε για το θέμα του Brexit τώρα. Το είχα στο μυαλό μου, αλλά μετά είχα αμφιβολίες. Ε, γιατί πρέπει να δούμε και το χρονικό διάστημα 2017-2019. Μέσα σε αυτό θα γίνει το Brexit. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για μια πιθανή μεταβατική περίοδο. Τέλος πάντων, είχα αμφιβολίες. Να το βάλω, αρχικά σκεφτόμουν στην έκθεση αλλά είμαι σίγουρη, ήμουν σίγουρη ότι κάποτε θα επανέλθει στην έκθεση ε, μέσω της κερκόπορτας των τροπολογιών. Το άφησα λιγάκι στον αέρα, ούτως ώστε μέσω των τροπολογιών να μιλήσω και για αυτό το θέμα, για τον Brexit δηλαδή. Ευχαριστώ. Προβλέπουμε ότι οι τροπολογίες θα κατεθούν στις 6 Νοεμβρίου τώρα, μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Θα, θα το συζητήσουμε στην Μπάτζα 22 Νοεμβρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμού στις 4 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2018. Κύριο, κύριε Βιώτη, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, Αλμαβίβα αυτό το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο μετεγκαθίσταται. Grazie, grazie, ehm, Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως και εδώ, έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Η Αλμαβίβα χαρακτηρίστηκε από την Ιταλική κυβέρνηση ως μια περίπτωση επιχείρησης που ε, θα κοστίσει για το Ιταλικό κράτος 5,5 εκατομμύρια, τα 3,5 θα πάνε από το Ταμείο. Μιλάμε για 1.646 ε, εργαζόμενους, 96% είναι γυναίκες, έτσι. Ε, μέχρι, που δούλευαν σε αυτό το κέντρο, το τηλεφωνικό κέντρο, μέχρι τα 55 ήταν η ηλικία τους. Έχουμε απίστευτη κρίση στον τομέα αυτό, των call center, των τηλεφωνικών κέντρων, ε, γιατί η Αλμαβίβα ήταν ένα τέτοιο τηλεφωνικό κέντρο. Στην Ιταλία, όπως και στην Ευρώπη, ε, προσπαθ... περνάνε από μια πολύ έντονη φάση αναδιάρθρωσης. Η Αλμαβίβα, στη συγκεκριμένη φάση, μείωσε το προσωπικό της κατά 46% και δυστυχώς δεν κατάφερε να υπάρξει συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους ικανοποιητική ούτω ώστε να ανταποκριθεί στι ανάγκε των εργαζομένων, που είναι κυρίω γυναίκε, όπω σα είπα. Η αρχική ε, χρηματοδότηση μέσω του ταμείου αυτού θα εξασφαλιστεί για να αποζημιωθούν ε, οι εργαζόμενοι. Και υποστήριξη για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ε, η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο στην Ιταλία ετοιμάζουν ένα νέο νόμο αρκετά ευνοϊκό για τους εργαζόμενους, ούτως ώστε να καθοριστούν οι σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην εταιρεία, ε, με ιδιαίτερη εστίαση ε, στους εργαζόμενους των call center, που μέχρι στιγμή δεν επωφελήθηκαν από ιδιαίτερα νομοσχέδια. Ε, στην πραγματικότητα δεν έχουν δείχτη ασφαλείας, δηλαδή νομοθετικής φύσεως. Γι' αυτό η Ιταλική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο κάνουν κάτι. Θα θυμάστε τι προθεσμίε. Ελπίζω να συζητηθεί αυτό το θέμα στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Του περιμένουν πάρα πολύ στην Ιταλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχουν ερωτήσεις. 17 Οκτωβρίου. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογίων 9 Νοεμβρίου η, προ... η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και τον ε, Νοέμβριο θα περάσει στην Ολομέλεια. Ο κ. Νόβακοφ. Youth Employment Initiative, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Το 2014, το πρώτο μου έτος στο Κοινοβούλιο, ήταν και η αρχή της ε, θητείας της Επιτροπής ε, Juncker. Μία από τις μεγάλες υποσχέσεις που ακούσαμε τότε ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι νέοι, στα πιο πολλά κράτη-μέλη. Νομίζω ότι έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση έκτοτε. Το έγγραφο που θα σας παρουσιάσω σήμερα έχει ως σκοπό να αποτυπώσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουμε σημειώσει. Παρά το γεγονός ότι καλύπτει τα όσα έχουν επιτευχθεί ως τώρα, εγώ προτιμώ να στρέφουμε πάντα στο μέλλον και όχι τόσο στο παρελθόν. Να μιλήσω δηλαδή για την περίοδο μετά το 2020 ό,τι αφορά την ε, ενίσχυση της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Έξι είναι θεωρώ τα βήματα για τις μελλοντικές μας εργασίες. Καταρχάς, ε, πιο πολλές επενδύσεις και πιο καλές επενδύσεις. Αυτό πρώτο. Επειδή υπάρχουν αποτελέσματα ήδη. Ναι, νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι πρωτοβουλίε για την απασχόληση των νέων και η εγγύηση για τους νέους είναι κάτι το οποίο προβάλλεται στα κρατη αν θέλετε, κατά του λαϊκισμού. 60.000 ε, νέοι στη χώρα μου και μόνο βρήκαν σταθερή δουλειά χάρη στο πρόγραμμα αυτό. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα κατά του προγράμματος. Το μέλλον, λοιπόν, θεωρώ είναι να πάρει άλλη κλίμακα το πρόγραμμα, να επενδυθούμε πιο, πιο πολλά και πιο αποτελεσματικά μέσα. Ύστερα, στρατηγικός σχεδιασμός. Να μην μετράμε μόνο τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται και να κάνουμε λογιστικά. Αλλά να δούμε τελικά πόσους βοηθάμε ουσιαστικά, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούμε και πόσο πιο λίγοι είναι οι νέοι που δεν έχουν κατάρτιση, εκπαίδευση. Απλοποιημένα, να τα πω τα πράγματα απλά δεν ε, μπορούμε να βρούμε οποιοδήποτε λόγο να κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζονται για τους νέους σε κάποιες περιπτώσεις έχει υπερβολικά αυστηρούς ε, όρους και προϋποθέσεις και προωθείται σε μέρη όπου δεν πηγαίνουν οι νέοι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό ως αλλαγή. Νομίζω ότι είναι εφικτό. Να αφήσουμε κατά μέρο περίπτωση διαδικασίε χρονοβόρε και εξαιρετικά μη φιλικέ προ τον χρήστη. Επίση, το πέμπτο βήμα το οποίο έχω γράψει, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και να προβάλλουμε καλύτερα τα αποτελέσματά μα. Γιατί πολλοί κόσμοι έχουν βρει δουλειά μέσω τη εγγύηση των νέων και όταν μιλάμε τελικά με αυτού, όταν του ρωτάμε πώ βρήκε δουλειά, τι έγινε, πιστεύουν ότι του βρήκε δουλειά ο υπουργό, ο δήμαρχο. Ε. Αλλά σε πολλέ περιπτώσει αγνοούν ότι τελικά η δουλειά οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε πιο πολλά για να εξηγήσουμε στον κόσμο το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και πώς ωφελεί τους νέους και πώς βελτιώνει τη ζωή τους. Θα προτιμούσα να ακούσω τη γνώμη των συναδέλφων και φυσικά η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή αν επιθυμείτε να καταθέσετε τροπολογίες, θα λάβω υπόψη όλες τις απόψεις. για να συνοψίσω για μένα η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν αποτελεί ένα τυχαίο αριθμητικό στοιχείο είναι ένα επιχείρημα, ένα χαρτί το οποίο θα πρέπει να παίξουμε στο τελευταίο 1,5 έτος του Κοινοβουλίου για να δείξουμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Θέλω να επεκταθεί, να ενηλικιωθεί, να πετύχει πιο πολλά, να πετύχει πιο πολλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι η βάση στην οποία βρισκόμαστε και επί της οποίας εργαζόμαστε είναι πολύ καλή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι όντω είναι θέμα προτεραιότητα αυτό, γιατί είναι ντροπή και όνειδο ενέργεια των νέων στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν δύο σκιώδει ε, εισηγητέ, τον κύριο Τενανό. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είχα προβλέψει να πω πολλά πράγματα, αλλά θα προσπαθήσω κι εγώ να, είμαι σύντομο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πράγματι, επί ουσία, συμφωνώ με τον κύριο Νοβακόφ σε πολλά. Συμφωνώ ως προς τη σημασία του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό να το επενθυμίζουμε ξανά και ξανά για τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, για την επικοινωνία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και αναφερθήκατε σε αυτά και πολύ καλώς. Στηρίζω την έκθεση. Τρία σχόλια έχω να διατυπώσω για τον κίνδυνο ενδεχομένως που υπάρχει να συγχωνευτούν οι διάφορες πηγές γιατί υπάρχουν διάφορες πηγές που μας έρχονται από παντού. Έχουμε το εργαλείο την εγγύηση για τους νέους, την πρωτοβουλία αυτή. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικών Εγγυήσεων, έχουμε το Σομαλή Λεγγύης, έχουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία ε, δεν πρέπει να χαθούν με τη συγχώνευση όταν τα βάζουμε όλα μαζί. Συμφωνώ ωστόσο με την απλούστευση. Δεν μπορούμε μονίμως και συνεχώς να έχουμε αξιολογήσεις προληπτικές και εκ των υστέρων, εξάντε και εξ post. Εκ των προτέρων σίγουρα πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να είναι αναπόσπαστη προϋπόθεση για να εγκριθεί ε, ένα έργο. Αν χρειάζεται χαρτούρα και γραφειοκρατία, Τια τεράστια για να εγκριθεί ένα έγκρο, τότε σίγουρα θα υπάρξει τη χαρτούρα και η γραφειοκρατία και μπορεί και να μην υπάρξει τίποτα μετά, να μην δοθεί συνέχεια. Τώρα, ε, για τις προϋποθέσεις εκ των υστέρων το αποτέλεσμα μετράει. Δηλαδή πόσοι νέοι τελικά βρήκαν δουλειά χάρη στο μηχανισμό. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο το θεμελιώδες για την αξιολόγηση εκ των υστέρων και αυτό πρέπει να προβληθεί. Επομένως, συμφωνώ αρκετά με το περιεχόμενο. Σίγουρα θα υποβάλω τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτών που σας εξέφρασα, αλλά δεν διστάνται και πολλοί απόψεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Ανελή, για παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει σημαντική οικονομική στήριξη στο πεδίο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και πρέπει να συνεχίσει να το πράττει αυξάνοντας το κονδύλι αυτό στον προϋπολογισμό. Η πρωτοβουλία για τους νέους θα πρέπει να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για μεταρρύθμιση και αλλαγή των πολιτικών στα κρατη και για καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους σε θέματα απασχόλησης και εκπαίδευσης. Αυτό πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο και με πιο μεγάλη ένταση στις χώρες μέλη που η ανεργία των νέων είναι εξαιρετικά υψηλή. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να γίνει ανταλλαγή από απόψεων για τις βέλτιστες πρακτικές και βέλτιστους τρόπους προσέγγισης της, ε, ε, του προβλήματος ε, της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Είναι μια κοινή πολιτική που μοιράζονται τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να παραμείνει τέτοια. Δηλαδή να το, όλα τα κράτη-μέλη το έχουν ιεραρχήσει ψηλά στον κατάλογο των πολιτικών τους προτεραιοτήτων. Όμως είναι και πρόκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραμένει ω πρόκληση δυστυχώ. Και τέλος να τονίσω ότι για να μειωθεί η ανεργία των νέων θα πρέπει τα κονδύλια να είναι στόχο προσιλωμένα, να είναι σωστά στόχοθετημένα... και οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να γίνουν αντικείμενο σύγκρισης για να δούμε εκεί ε, όπου υπάρχει η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το συμπέρασμα είναι ότι πολλά ακόμα μένει να γίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος άλλος θέλει το λόγο, κανείς. Κύριε Νοβάκοφ, δύο λόγια θα ήθελα να πω. Η Επιτροπή την 5η 5 Οκτωβρίου δημοσίευσε ένα σχέδιο που είναι πρόταση συστάσεων προς το Συμβούλιο για να αναπτυχθεί στην Ευρώπη ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μαθητεία, το οποίο να είναι αποτελεσματικό και ποιοτικό. Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το εργαλείο, θα μπορούσε κανείς αυτό το εργαλείο να το ενισχύσει για να ενισχύσει τη μαθητεία γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αυτή την παράδοση ε, της μαθητείας και του ισχυρού πλαισίου μέσα σε αυτήν έχουν ένα ποσοστό απασχολησιμότητας των νέων τους πολύ ψηλότερο από τις υπόλοιπες. Άρα δεν μπορεί να βρει αυτό το σχέδιο τη θέση του στην πρωτοβουλία για το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μαθητεία. Έχετε το λόγο. Πράγματι θα μπορούσε. Κύριος Νοβάρτης θέλει να πάρει το λόγο. Μακάρι να χάναν τη σημασία τους σύν το χρόνο αυτά τα, αυτοί οι μηχανισμοί υπέρ της απασχόλησης των νέων. Αλλά φοβάμαι πως όχι, γιατί θα αλλάξει και η φύση της οικονομίας. Αυτά, αυτοί οι μηχανισμοί απλώς θα πρέπει να προσαρμοστούν. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Για, μπορεί να έχουμε μία μονόπαντη προσέγγιση για τα πάντα. Το βασικό είναι να δούμε τα καλύτερα συστήματα και να φτιάξουμε τελικά μία δέσμη κριτηρίων που είναι τα καλύτερα κριτήρια για να τα αξιολογούμε όλα αυτά. Να μάθουμε δηλαδή και όταν μαθαίνουμε να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν ανάγκες ε, αλλαγής, προσαρμαστής, ανάπτυξη αξιών, να καταλάβουμε πώς μπορούμε να υποφεληθούμε καλύτερα από αυτά τα συστήματα, αλλά θα πρέπει να το να το αποδείξουμε και αυτό το πράγμα σύν και να προσαρμόζουμε αυτούς τους μηχανισμούς στις, α, ε, στις αλλαγές της, οικονομίας μας. Ο εισηγητής θα καταλήξει τώρα σε κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Το πιο προβληματικό, το πιο δύσκολο πράγμα με την ενεργεία των νέων είναι ότι μία προσέγγιση, πιο ας πούμε για την Ελλάδα ή την Ισπανία, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ούτε στην Σουηδία, ούτε στη Φιλανδία, ούτε στο Βέλγιο, ας πούμε. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να αφήσουμε τις τοπικές αρχές και τις εθνικές αρχές να βρουν την καλύτερη προσέγγιση για το κοινό στόχο, το κοινό παύλα στόχο γιατί αν έχουμε ένα πρότυπο για, τα, όλους, σε κάποια κράτη-μέλη, σε κάποιες περιοχές, λόγω της φύσης του προβλήματος και λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι νέοι, 9 στις 10 περιπτώσεις θα είναι τέλεια τα πράγματα. Αλλά σε ένα άλλο κράτος μέλος, λόγω του ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα, γιατί η κουλτούρα και το εκπαιδευτικό σύστημα ή γενικά διάφορα άλλα πράγματα είναι αλλιώτικα, δεν θα λειτουργήσει. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι σωστό. Καλή είναι η προσέγγιση αυτή, αλλά όχι, δεν μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο πράγμα και στα 27 κράτη-μέλη. Εν γέννη θα παίξει θετικό ρόλο και θα βοηθήσει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο διάφορους νέους. Το πρόβλημα βρίσκεται σε διάφορα επίπεδα. Αν δεν βρούμε μια βιώσιμη λύση τώρα, σε πέντε χρόνια δεν θα έχουμε απλώς ανεργία. Θα φύγουν οι νέοι μας προς άλλες περιοχές του πλανήτη, θα επηρεαστεί η Ευρώπη, δεν θα έχουμε πια νέους επιστήμονες, δεν θα έχουμε νέους καλλιτέχνες, δεν θα έχουμε νέα ταλέντα στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, κλπ. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει και θα πρέπει να πέσει θύμα περικοπών του προϋπολογισμού. Δεν θα πρέπει να πάρουμε λεφτά από εκεί για να χρηματοδοτήσουμε άλλα προγράμματα, να αντιμετωπίσουμε άλλες κρίσεις. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να δώσουμε ασφάλεια στον κόσμο. Ναι, και για τα θέματα των προσφύγων, για τον έλεγχο των συνόρων κτλ. Αλλά να κρατήσουμε και αυτή την προτεραιότητα για την ανεργία των νέων και το πώς αντιμετωπίσουμε και αν το κάνουμε αυτό θα το εκτιμήσουν οι σημερινοί νέοι και οι επόμενες γενιές. Βλέπουμε ότι τα ταμεία συνοχής δεν χρησιμοποιούνται. Θα επιστρέψουμε 7 δισεκατομμύρια στα κράτη-μέλη. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η επένδυση στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων μέσω της μαθητείας, ας πούμε. Είναι μια επένδυση καλή για το μέλλον, για να διευκολύνει την απασχολησιμότητα των νέων πατού στην Ευρώπη. Έρθω σε επαφή και διμερώς μαζί σας για να τα συζητήσουμε αυτά. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί φέτος ε, θα έχουμε 7 δις ε, υπόλοιπο που θα επιστρέφουν στα κράτη-μέλη, όπως είπατε. Αλλά να με θυμηθείτε, σε ένα χρόνο θα έχουμε τόσες πολλές, τόσο πολλά αιτήματα για πληρωμές που θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί συμπεριφέρονται έτσι τα κράτη-μέλη και είναι δύσκολο επίσης να ζητάμε πιο πολλά γιατί ακόμα και αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας τώρα δεν αξιοποιούνται πλήρως. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί έχει πως και η κατάσταση της πολιτικής συνοχής στην παρούσα φάση. Αλλά νομίζω ότι και η εγγύηση για τους νέους και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μπορεί να συνάδουν με την πολιτική συνοχή και τα τελευταία ταμεία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας πω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να κατευθούν το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου πέντε το απόγευμα και στις 22 Νοεμβρίου έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, 4 Σεπτεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Καθελήν Αρμόδια, που είναι η Επιτροπή Απασχόλησης, το Δεκέμβριο θα ψηφιστεί το θέμα στην Ολομέλεια. Και περνάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης το οποίο το, για τον οποίο υπεύθυνο είναι ο Γιάνν Σκέιερ, ο οποίος είναι υπεύθυνο ε, επίσης εισηγητής ε, και για τις ε, εξωτερικές υπηρεσίες Τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα συστήματα IT. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω. έχουμε το highlight στο τέλο τη βραδιά. με, γενικές, ε, με μια γενική αξιολόγηση και σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του Ιωλίζα, ο βασικός κανονισμός λοιπόν ε, της ε, υπηρεσίας αυτής ε, περνάει από αναθεώρηση και αυτό έχει να κάνει με τους πολιτικούς τομείς που σε εμά το Κοινοβούλιο κοιτάει η Επιτροπή για τα δικαιώματα του πολίτη. Η Αγιουλίζα λοιπόν διαθέτει μεγάλες βάσεις δεδομένων για την τεχνική εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων γύρω Schengen, European Travel Innovation, Information Authorization System. Έχει έδρα στο Τάλιν, στην Εσθονία, αλλά έχουν και να γραφτεί στο Στρασβούργο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό όπου έχουν ε, τους υπολογιστές τους και τα backup τους γίνεται στην Αυστρία. Πραγματικά λοιπόν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταναμημένη σε διάφορα κρατημέλη. Από πλευρά σε προπολογισμού δεν έχουμε πολλά να πούμε. Σε ό,τι αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρώτη παράγραφο ε, έχει να κάνει με την άμεση ενίσχυση σε εξαιρετικέ καταστάσει έκτακτη ανάγκη. Ε, το Ιουλίζα, λοιπόν, έχει και ασχολείται με το θέμα τη κατανομή του κόστου. Η υπηρεσία υποτίθεται ότι αναλαμβάνει το επιπρόσθετο κόστο για να μην επιβαρύνει το κράτο μέλος. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει σωστός προπολογισμό για την υπηρεσία. αν θέλει να συνεργαστεί στενά μία ομάδα έξι κρατών μελών μπορεί να επικληθεί τη βοήθεια της υπηρεσίας στην τροπολογία υπεριθμών 4. Ζητούμε κάτι το οποίο ζητάμε παντού όπου χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να διορίσει ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας και αυτό ανταποκρίνεται στη θεσμική συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων για τις εξωτερικές αυτές υπηρεσίες. Πέμπτη τροπολογία. Θα την αναγνωρίσετε. Η μεταφραστική υπηρεσία της ε, Γιουλίζα είναι υπερφορτωμένη, δεν έχει επαρκές προσωπικό. Άρα οι μεταφραστικές αυτές υπηρεσίες θα πρέπει να περνούν από εξωτερική ανάθεση, αν αυτό απαιτείται. Το Διοικητικό Συμβουλίο θα πρέπει να περνάει από αξιολόγηση, αναφέρεται αυτό, και στην τροπολογία υπαριθμών 7 δεν έχουμε ακόμα οριστική εκτίμηση όλων των τροπολογιών, των τροποποιήσεων που γίνεται στο βασικό αυτοκανονισμό. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την εξετάση αυτή. Εξετάζουμε ακόμα το ρόλο του διευθυντή και το θέμα της κατανομής του κόστους ε, σε ό,τι αφορά συμφωνίες συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές εξωτερικές υπηρεσίες στις 12 Οκτωβρίου την επόμενη Πέμπτη είναι η προθεσμία για την κατάθεση των... Ε, ελπίζω μέχρι τότε να το έχουμε διευκρινίσει το θέμα αυτό με το γραφείο μου. Επίσης, ε, τονίζουμε το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας, αλλά το βγάζουμε και το βάζουμε μάλλον σε αγγίλες, γιατί δεν έχει επιπτώσεις καθόλου στον προπολογισμό. Αυτό φυσικά να το συζητήσουν οι συνάδελφοι. Από τη Λίμπε, εμάς δεν μας επηρεάζει καθόλου από πλευρά τη Επιτροπή μα. Δεν έχει δημοσιονομικέ επιπτώσει και άρα δεν θέλησα να τοποθετηθώ από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Μας διαφωτίσατε. Οι σκιώδεις εισηγητέ θέλουν να πάρουν το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Δεν θέλουν να παρέμβουν έχουν εμπιστοσύνη στον εισηγητή που ε, συμπεριέλαβε με μεγάλη ακρίβεια τα σημεία που τους ανησυχούν. Καταληκτική προθεσμία τροπολογιών 12 το μεσημέρι μεθαύριο, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 22-23 Νοεμβρίου. Άρα, δεν σας δίνω το λόγο για να αντιδράσετε στις παρατηρήσεις των σκιωδών εισηγητών, γιατί δεν παρατήρησαν τίποτα και δεν έχετε τίποτα να προσθέσετε σε αυτά που μόλις τώρα μας είπατε. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας διαφωτίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι και εγώ μπορώ να είμαι πολύ σύντομος να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης εξετάσαμε προσεκτικά τις οκτώ προτινόμενες τροπολογίες. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με καμία από αυτές, ουσιαστικό. Βεβαίως, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θα προτιμούσαμε την αρχική διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αυτό δεν σας εκπλήσει ποτέ νομίζω. Σε άλλες τροπολογίες, με άλλες συμφωνούμε απολύτως, όπως η 3 και η 8. Δεν υπάρχουν προβλήματα βασικά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Καλώ, λέει ο πρόεδρο. Η συνέχεια προμηνύεται πολύ θετική, κύριε εισηγητά. Θα έχετε τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά λοιπόν. Υπό τα διάφορα. Ποιος θέλει να θέσει κάτι υπό τα διάφορα. Τίποτα. Κανείς. Πολύ ωραία. Λίγη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Και ε, εκφράζω την, ε, θερμές μου ευχαριστίες για όσους από εσά έμειναν μέχρι τέλους. Ε, λήξη της συνεδρίασης.